Hyvää huomenta. Voimme aloittaa kokouksen. Καλημέρα. Νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση. Δεν έχουμε τόσο πολλούς συναδελφούς σήμερα εδώ μαζί μας ε, όσους είχαμε χθες ε, όταν συζητούσαμε δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε ενδιαφέροντα σημαίες στην ημερήσια διάταξή μας. Και γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Έχουν περάσει 20 χρόνια από κάποια συγκεκριμένα συμβάντα στην Κίνα και νομίζω πως θα πρέπει να τιμηθούμε αυτή την ημερομηνία και βέβαια αυτή ακριβώς η επέτειος ε, έχει οδηγήσει στη λήψη πολλών μέτρων ασφαλείας ενώ λήφθηκαν και ειδικά μέτρα περιορισμού σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο ε, πράγμα βέβαια το οποίο είναι ανησυχητικό για μας. Ε, πάρα πολλοί ακτιβιστές και υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συλλήφθησαν και τους ε, ζητήθηκε να εγκαταλείψουν το Πεκίνο ενώ κάποιοι απήχθησαν. Ε, και όσοι είχαν ε, μετακινηθεί εκεί ούτως ώστε να παραπονεθούν στις αρχές τους ζητήθηκε να επιστρέψουν πίσω στις περιοχές τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό και θα πρέπει να επιστήσουμε με σοβαρό τρόπο την προσοχή της ε, Κίνας ώστε να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Είναι θλιβερό το ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει την 20η επέτειο. Το επόμενο σημείο είναι η ώρα των ερωτήσεων και έχουμε ένα κατάλογο από πέντε ερωτήσεις και τις ε, απαντήσεις της Επιτροπής σε αυτές. Ε, Η πρώτη ερώτηση είχε κατεθεί από την Μπάρβαρα Λόχμπιλερ και αφορά την ε, παιδική εργασία. Η κυρία Λόχ ε, Μπίλερ ε, θέτει ένα ερώτημα σχετικά με μια έκθεση την οποία έχει υποσχεθεί να καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είχε δεσμευτεί να μας υποβάλει τα πορίσματα της σχετικής έρευνάς της και την έκθεσή της πριν από το καλοκαίρι. Υπήρξε λοιπόν μια καθυστέρηση εδώ και η κυρία Λόχμπιλερ ζητάει να μάθει γιατί σημαίνει αυτή η καθυστέρηση και ζητεί μια α, κατάλληλη έκθεση, επίσημη έκθεση και όχι μόνο τα ανεπίσημα έγγραφα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ε, τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιος θα πάρει το λόγο, κύριο Στήμανς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, επικεφαλής της σχετικής ε, μονάδας ε, Digitrade και είμαστε η αρμόδια μονάδα για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης με βάση και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2008. Ε, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή αυτής της έκθεσης ενώ και η ακριβής μορφή που θα λάβει αυτή η έκθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς αυτή θα ακολουθήσει την ουσία της, το περιεχόμενό της. Δηλαδή όταν θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο θα αποφασίσουμε τι μορφή θα δώσουμε σε αυτή την έκθεση. Και βέβαια ε, προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας και το νέο θεσμικό περιβάλλον, δηλαδή το νέο ε, κοινοβούλιο ε, και τις διαβουλές που μπορούμε να έχουμε με τα μέλη του κοινοβουλίου για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα μας επιτρέψει να δώσουμε ε, έναρξη μας περαιτέρω συζήτηση και όχι απλά να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα ή κάποιες συστάσεις. Έχουμε προχωρήσει αρκετά με την εκπόνηση αυτού του σχεδίου και ελπίζουμε πως θα, και αναμένουμε πως θα έχει οριστικοποιηθεί ε, στο εγγύς μέλλον, σίγουρα μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας συντολής, της τρέχουσας δηλαδή Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παιδική εργασία, ώστε να δούμε ποια είναι τα περαιτέρω μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για την ε, ακόμα πιο αυξημένη καταπολέμηση τη παιδική εργασία. Ελπίζω να σας κάλυψα με τι απαντήσει μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα ήθελε να πάρει το λόγο ε, Λόχμπιλερ για να θέσει κάποιο περαιτέρω ερώτημα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, μια διευκρίνηση θα ήθελα να ζητήσω γιατί θα πρέπει να αποφασίσουμε εκ νέου ποια μορφή θα λάβει τελικά αυτή η έκθεση. Ε, νομίζω πως είχαμε τονίσει πως είναι απαραίτητο να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης και να μην αποτελέσει απλώς μια άτυπη ενημέρωση. Ε, ενδεχομένως να κάνω κάποιο λάθος, ε, νομίζω να μην έχω καταλάβει ακριβώς. Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε να μας ε, διευκρινίσετε λίγο, να μας δώσετε μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την δεύτερη ερώτηση. Ε, ζητώ συγγνώμη αν δεν ήμουν σαφή για την πρώτη μου παρέμβαση. Η μορφή λοιπόν που θα λάβει, εάν θα υπάρξει ένα working paper, δηλαδή έγγραφο εργασία ή ανακοίνωση οτιδήποτε άλλο, θα εξαρτηθεί από την ουσία του της έκθεσης δηλαδή. Εάν είναι αναλυτικό το έγγραφο, ε, τότε ε, η πιο ενδεδειγμένη μορφή είναι να αποτελέσει έγγραφο εργασία. Εάν όμω έχουμε συγκεκριμένε συστάσει σε ό,τι αφορά τη χάραξη τη πολιτική, τότε θα πρέπει να αποτελέσει ανακοίνωση κάτι άλλο. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία είναι περισσότερο γραφειοκρατικά, τα οποία ορίζουν την μορφή, για παράδειγμα ο αριθμό των σελίδων και ούτω καθεξής. Ε, αλλά ε, το κύριο κριτήριο ε, για τη μορφή που θα επιλέξουμε να έχει αυτή η έκθεση θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο, από την ουσία της. Ελπίζω να σας κάλυψα τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ναι, νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Ελπίζουμε λοιπόν να περσότερα. περισσότερα Επόμενη ερώτηση από Κριστιαν Νταν Μπρέντα σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μιαμάρ και τι ε, ερχόμενε κοινοβουλευτικέ εκλογέ στη χώρα ε, του χρόνου. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως οι εν λόγω εκλογές θα είναι ελεύθερες και δίκαιες. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ποια μέτρα ενδεχομένω θα λάβει το ε, στρατιωτική χούντα στη χώρα την ενόψη αυτών των εκλογών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Σήμερα ακόμα δεν υπάρχει εκλογικός νόμος που να καθορίζει την κατάσταση για τις εκλογές που προβλέπονται το 2010. Ούτε για τους μελλοντικού υποψηφίους, ούτε και για τα πολιτικά κόμματα. Και γι' αυτό είναι δύσκολο, προς το παρόν τουλάχιστον, ε, να ξέρουμε κατά πόσο ο μελλοντικό εκλογικό νόμο θα είναι ιδιαίτερα περιοριστικό ή όχι. Συνεπώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δικιά τη την πλευρά δεν θέλησε να εκφραστεί όσον αφορά τι συνθήκε συμμετοχή στι εκλογέ αυτέ. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιμόνω ζητάει από τις αρχές να φροντίσουν ώστε οι εκλογές του 2010 να επιτρέψουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Στο ίδιο πνεύμα δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει διάλογο με τις αρχές προκειμένου να ελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και για να στηριχθεί η ανάπτυξη και η κοινωνία των πολιτών εκεί. Ευχαρίστω από εκεί και πέρα να απαντήσω σε συμπληρωματικές ερωτήσεις εφόσον έχετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Σίγουρα ο κύριος ε, Πρέντα θα έχει συμπληρωματική ερώτηση, έτσι δεν είναι. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η μόνη ερώτησή μου είναι εξή. Βλέπετε με εκπλήσει λίγο η αξιολόγηση αυτή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Εφόσον το Σύνταγμα της Βερμανίας περιορίζει ήδη το δικαίωμα ε, κατάθεσης υποψηφιότητος για όσους είναι παντρεμένοι με ξένους. Καταλαβαίνετε, υπάρχει περίπτωση ο εκλογικός νόμος να αντιβαίνει στο Σύνταγμα και να επιτρέπει την ελεύθερη συμμετοχή όλων προκειμένου να υποβάλουν υποψηφιότητα. Θα ήταν τεράστια καινοτομία αυτή. Το Σύνταγμα περιορίζει το δικαίωμα και ο εκλογικό νόμο να επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία. Ε, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τέλο πάντων, οπότε αυτό είχα να πω. Καλώς. Το συνταγματικό θέμα είναι ένα θέμα στο οποίο σίγουρα θα μπορεί να σας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι το Σύνταγμα προβλέπει απαγόρευση μεταξύ άλλων όσων είναι παντρεμένοι με ξένους να υποβάλουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν ως ηγέτες του κράτους. Αυτό είναι ο περιορισμός που υπάρχει σήμερα. Ο κύριος Πρεντά αναφέρεται στην κυρία Σουτσή φαντάζομαι. Προς το παρόν, προς το παρόν έτσι. Δεν υπάρχει νόμος που θα μπορούσε να υπαγορεύσει να είναι υποψήφια ή να ψηφίσει. Προς το παρόν. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εννοείται ότι σίγουρα θα ξαναμπεί στην ημερήσια διάταξη Μιαμάρ με τις εκλογές που έρχονται. Η κυρία Μπρεπούλς τώρα έχει ρωτήσει για την κατάσταση όσον αφορά τα παιδιά στην Παλαιστίνη. Αναφέρεται σε διάφορες συμβάσεις, συνθήκες και συμφωνίες προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού. Μπορείτε παρακαλώ να απαντήσετε που βγάζει Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και χτες λιγάκι το θίξαμε αυτό το ζήτημα. Επιτρέψτε μου να σας πω τα εξής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται απόλυτα τις ανησυχίες που εκφράζει η αξιότιμη Ευρωβουλευτής. Όσον αφορά την κατάσταση παιδιών Παλαιστινίων στις φυλακές του Ισραήλ. Αυτό είναι ένα θέμα στο κέντρο των συζητήσεων που έχουμε με τους Ισραηλινούς σε διάφορα επίπεδα και ιδιαίτερα στα πλαίσια της άτυπης ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνεδρίασε για τελευταία φορά στις 3 Σεπτεμβρίου. Εκεί θίξαμε για άλλη μια φορά αυτό το ζήτημα. Τώρα αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει πως καθορίζοντας την ηλικία κράτησης στα 16 χρόνια, αυτό είναι κάτι που δεν ευθυγραμμίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών. Είναι επίσης κάτι διαφορετικό από την τρέχουσα νομική κατάσταση στο Ισραήλ που μιλάει για τα 18 χρόνια, ότι δηλαδή είναι κάποιος ανήλικος μέχρι τα 18 του. Εμείς θεωρούμε ότι τα παιδιά αυτά που βρίσκονται σε κράτηση στο Ισραήλ, είτε διοικητικά είτε κανονικά βάσει του ποινικού δικαίου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε η κατάσταση να συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Οι Ισραηλινοί εξήγησαν ότι στις 29 Ιουλίου οι στρατιωτικοί από το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη προσπάθησαν να διαθετήσουν την κατάσταση όσον αφορά τους ανήλικους και το Ισραήλ τώρα έχει φροντίσει να υπάρχει δική δικαιοδοσία για τα παιδιά, δική νομολογία δηλαδή, που αρχίζει να ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2009. Πάντως, οι επικρίσεις παραμένουν παρόλα αυτά. Κυρίως παιδιά Παλαιστίνοι εξακολουθούν να βρίσκονται ε, υποκράτηση χωρίς δικηγόρο, χωρίς την παρουσία δικών τους, γονιών τους, συγγενών τους. Υπάρχει και η Επιτροπή για τα Βασανιστήρια που είπε ότι έπρεπε να μαγνητοσκοπούνται οι ανακρίσεις που γίνονται. Δεν δόθηκε όμως συνέχεια σε αυτό. Από όσο γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως τέλη Ιουλίου, 342 παιδιά, ανήλικοι δηλαδή Παλαιστίνοι, κρατούνται από το Ισραήλ. 42 σήμερα, 12 έως 15 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που το θίγουμε ξανά και ξανά. Επίσης πρέπει εδώ να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο γίνεται για την παρουσία παιδιά σε ζώνες όπου υπάρχουν συγκρούσεις. Ένας από τους στόχους των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών λοιπόν είναι η προστασία αυτών των παιδιών και έτσι προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή με τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών μας ε, στην περιοχή ώστε τοπικά να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν συνεργαζόμαστε και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Παλαιστίνη για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε τις εκκλήσεις μας προς το Ισραήλ να φροντίσει να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πρέπουλ σίγουρα θέλει να ρωτήσει κάτι ακόμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση που μας έδωσε και χτες εδώ και κλεισμένο το θυρών είχαμε συζήτηση για αυτό το θέμα το συζητήσαμε, αλλά παραμένουν οι ερωτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για την άτυπη ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χτες ενημερωθήκαμε σχετικά. Τώρα, διαβάζω στο ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο πέρυσι ότι στο Βούλιο με το Ισραήλ αποφασίστηκε η ομάδα αυτή εργασίας να αντικατασταθεί από ε, μία Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά χτες ακούσαμε ότι δεν έχει δοθεί συνέχεια σε αυτό. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Και ο πολιτικός διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ ε, προχωράει. Αυτή η υποεπιτροπή θα φτιαχτεί ποτέ. Έπειτα στο ίδιο ψήφισμα του Κοινοβουλίου το περσινό Σε σχέση με τις διοικητικές κρατήσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται, χαίρομαι που είπε και η Επιτροπή ότι υπάρχουν, τον τελευταίο χρόνο δεν έχουμε δει καμία πρόοδο. Αντίθετα, τα παιδιά εξακολουθούν να κρατούνται κάτω από τους ίδιους κανόνες όπως και οι ενήλικοι. Οπότε λοιπόν θέλω να ξέρω πώς είναι δυνατόν να ξεφεύγουν από τους κανόνες Ισραηλινοί με αυτόν τον τρόπο και να διώκονται και να κρατούνται πολίτες χωρίς την παρουσία δικηγόρου, χωρίς την παρουσία συγγενών τους, χωρίς μαγνητοσκόπηση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, για μήνες, χωρίς να γίνεται δίκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να κάνει περισσότερα γι' αυτό. Όλα αυτά παραβιάζουν κάθε είδους δίκαιο. Πρέπει να κάνουν λοιπόν ό,τι μπορούν, ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να διορθωθεί η κατάσταση. Και εμείς από το Κοινοβούλιο ίσως θα μπορούσα να ρωτήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής μας Μήπως μπορούμε να, ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπενθυμίσει το ψήφισμα που ανέκρινε πέρυσι το Κοινοβούλιο, να το υπενθυμίσει στις Ισραηλινές αρχές μια που δεν έχουν κάνει τίποτα για τη βελτίωση της κατάστασης. Ευχαριστούμε, κύριε Μπρέπουλς. Σωστά. Καλά κάνετε και μας υπενθυμίζετε και υπογραμμίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αλλά ίσως η Επιτροπή, ο κύριος δεν μπορεί ακόμα να απαντήσει. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, δηλαδή τη δημιουργία αυτή της υποεπιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω το πρότεινε στο Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν το δέχτηκε. Και το Ισραήλ προτίμησε μια προσαρμογή των δομών των επιτροπών που υπάρχουν βάσει των διμερών συμφωνιών. Ιδιαίτερα στα πλαίσια διαπραγματεύσεων για ενισχυμένες σχέσεις. Αλλά, όπως γνωρίζετε, αυτή η αναβάθμιση σχέσεων έχει σταματήσει, έχει διακοπεί μετά το πόλεμο στην Γάζα τον Ιανουάριο. Συνεπώς, προς το παρόν, έχουμε αυτή την άτυπη ομάδα εργασίας μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που, όπως σας είπα, συνεδρίασε πρόσφατα. Πάντως, θέλω να επαναλάβω την ε, θέση μου όσον αφορά την κράτηση παιδιών στις Ισραηλινές φυλακές και όσον αφορά τις ποινικέ διαδικασίες και ακόμη και τη διοικητική κράτηση, ότι αυτό το θέμα έχει τεθεί στους Ισραηλινούς. Και είμαστε έτοιμοι να το θέσουμε και πάλι σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε επίπεδο αυτής της άτυπης ομάδας εργασίας, αλλά και υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης που έχουμε με το Ισραήλ. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο φυσικά πρέπει να αποφασίσει τι συνέχεια θα δώσει, τι δράσει θα αναλάβει προς ε, το Ισραήλ. Πάντως θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι και συζήτηση 14 Μαου του 2009 σε επίπεδο ΙΕ, η Αρμόδια Επιτροπή για τα Βασανιστήρια, που εκφράζει πάντα ανησυχίες για το γεγονός ότι ανήλικοι Παλαιστίνοι κρατούνται και ανακρίνονται στο Ισραήλ τη απουσία δικηγόρου ή της οικογένειάς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επανέλευε τις ανησυχίες της για τις υπόνοιες που ακούγονται για 700 παιδιά ετησίως τα οποία δικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια. 95% των περιπτώσεων αυτών βασίζονται σε ομολογίες ε, που ουσιαστικά με το ζόρι πήρανε από τα παιδιά αυτά. Είπαμε ότι θέλουμε νομολογία ειδικά για τα παιδιά και κανονικά αρχίζει να ισχύει από το Σεπτέμβριο φέτος. Καταλαβαίνετε είναι πολύ πρόσφατο, οπότε ακόμα δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί, αλλά πάντως στις, στα τέλη αυτής της χρονιάς, αρχές της επόμενης, θα έχουμε περισσότερες ε, πληροφορίες όσον αφορά τους ειδικού νόμους που θα αφορούν τις ε, κρατήσεις και τις διώξεις ανηλίκων. Είμαστε πάντως αποφασισμένοι να το θίγουμε ξανά και ξανά το θέμα σε κάθε επίπεδο με τις Ισραηλινές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κατάσταση για την οποία ρώτησε η κυρία Μέιπορς είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για το ότι υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή συμφωνιών και ψηφισμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να τα παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Τέταρτη ερώτηση, David Martin. Είναι κάπως ε, γενικά διατυπωμένη σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Κρίστον Φίσνερ. Είμαι υπεύθυνο για θέματα Κολομβία, desk officer. Πρέπει να έχουμε κατά νου από πού ποια είναι η προηγούμενη ιστορία. Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε πολλέ προσπάθειε να ενισχύσει το κράτο δικαίου στη χώρα. Υπήρχαν, υπήρχε βία εκ μέρου ε, των κυκλωμάτων ναρκωτικών, ανταρτών και άλλων παράνομων ομάδων. Εν μέρη πέτυχαν αυτές οι προσπάθειες και οι δείκτες της γενικής ασφάλειας βελτιώθηκαν. Σε μερικά μέρη πάρα πολύ. Στα ανθρώπινα δικαιώματα και εκεί είχαμε βελτίωση. Γι' αυτό η Ένωση κατ' επανάληψη υποστήριξε την πολιτική αυτή και στα πορίσματα του 2007 του Συμβουλίου Βέβαια, δεν τους υποστηρίζουμε και δεν τους βοηθάμε ανεφόρον. Υπάρχουν πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία που μας ανησυχούν πολύ, όπως πρόσφατες εκθέσεις από τον ειδικό εισηγητή των ΗΕ για τους ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εισηγητής για τους ε, ηθαγενείς Γι' αυτό είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη και στο διάλογο που έχουμε την Κολομβία, όλα αυτά για να έχουμε περαιτέρω πρόοδο. Για το διάλογο, πέραν των διαφόρων διεθνών πλαισίων που υπάρχουν, Συμβούλιο Ηνωμένων Εθνών κλπ. Η αναθεώρηση για την Κολομβία έγινε, η ανασκόπηση μάλλον έγινε τον περασμένο μήνα. Πριν από μερικού μήνε συναισθήθηκε μια διμερή ομάδα για διάλογο με την Κολομβία, πρώτη συνάντηση τον Αύγουστο, και η δεύτερη συνάντηση θα γίνει σε μερικές εβδομάδες. Εκεί είναι ένα βήμα όπου σκοπεύουμε <clears throat> να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και εμπειρίες και να δίνουμε και στοιχεία για τεχνική συνεργασία. Ελπίζουμε αυτό να οδηγήσει σε συγκεκριμένη πρόοδο. Και στον πολιτικό διάλογο, στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, με δράσεις ad hoc και εκεί τίθεται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρεμβάσεις. Συστηματικά ζητάμε από την Κολομβία να προστατεύσει τις ε, ευπαθείς ομάδες που είναι και οι προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πολλές φορές υφίστανται επιθέσεις εκπροσώπους ε, από συνδικαλιστικές οργανώσεις θύματα δολοφονιών έξω δικαστικές παράνομες φυσικά εκτελέσεις εκ μέρους των στρατιωτικών, όπως έγινε πέρυσι. Όλα αυτά πρέπει να ανακρίνονται γρήγορα και οι δράστες να τιμωρούνται. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μετράνε και στην συνεργασία μας και στα διμερή προγράμματα. Στα εργαστήρια ειρήνης, όπως τα λέμε στην Κολομβία, Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα στο θέμα της δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της ετοιμορρησίας. Ένα όλο πρόγραμμα για σταθερότητα, για βοήθεια των θυμάτων του δικαστικού συστήματος και άλλα προγράμματα για θύματα, για τις μειονότητες, για τους ε, ντόπιους ηθαγενείς με βάση το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλα αυτά θα συνεχιστούν με ψηλή προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την απάντησή της. Χαίρομαι που κρατάνε ψηλά στην ημερήσια διάδειξη των ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά πολύ φυσικαστική δεν βρήκα την απάντηση. Αληθεύει ότι πρόσφατα η Κολομβία βολτίζει το νομικό τη σύστημα σχετικά με τις καταχρήσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Σε μια χώρα όπω η Κολομβία κανένα δεν είναι απολύτω ασφαλή, αλλά τα στοιχεία μα δείχνουν ότι οι συνδικαλιστές και οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δολοφονούνται και δεν γίνεται ανάκριση από την κυβέρνηση. Και όπως είπατε μπορεί να έχουν γίνει και με εντολή της κυβέρνησης. Αυτό είναι παράδεκτο. Η Κολομβία υποφελείται από το εμπορικό σχήμα GSP συν της Ένωσης, σύστημα γενικημένων προτιμήσεων και όπως ξέρετε εκεί μέσα προβλέπεται η τήρηση των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν το κάνει αυτό η Κολομβία. Να αποσύρουμε αυτή την, αυτού του είδους τη συνεργασία των γενικημένων προτιμήσεων συν με την Κολομβία μέχρι ότου και, και να το μελετήσει το, το θέμα αυτό η Κομισιόν κατά πόσον πρέπει ή όχι να επανέλθουμε. Πρόεδρος. Η ερώτηση σχετικά με την χρήση των εργαλείων εμπορικής πολιτικής που θα ήταν κατάλληλα προς χρήση στην περίπτωση αυτή. Αυτή ήταν η ερώτηση. Η Κομισιόν παρακαλώ να απαντήσει. Απάντηση. Ευχαριστώ. Δεν εφησυχάζομαι. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία είναι δεινή. Τώρα ο βαθμός ατιμορρησίας. Η κληρονομιά των εσωτερικών συγκρούσεων στην Κολομβία είναι τεράστια. Και αυτό δεν αφορά μόνο οι ευπαθεί ομάδε όσον αφορά υπερασπιστέ, ακτιβιστέ, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικαλιστέ κλπ. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλέ δολοφονίε. Και ο βαθμό ατιμορρησία είναι πάνω από το 90%. Αυτό που έχει σημασία ποια είναι η τάση. Υπάρχουν όλο και περισσότερε καταδίκες, αν και το ποσοστό είναι χαμηλό. Ένα από του στόχου μα στα πλαίσια τη συνεργασία είναι να υποστηριχθεί ο δικαστικός τομέας, να αυξηθεί το ποσοστό καταδικών. Πιέζουμε την κυβέρνηση και προληπτικά να πάρει μέτρα. Παραδείγματος χάρη στα προγράμματα προστασίας για τις ευπαφείς ομάδες. Και εδώ μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Αυτοί που είναι υπό την επίσημη προστασία Ούτε μία δολοφονία δεν είχαμε σε αυτή την ομάδα. Θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση, να συζητάμε με την κυβέρνηση τι μπορούμε να κάνουμε και από κοινού για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την Κομισιόν. Πέμπτη ερώτηση. Ο αντιπρόεδρος κύριος Κάζακ Ερωτά για το στρατόπεδο Άσραφ στο Ιράκ και την κατάσταση εκεί. Πολύ ανησυχητική κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Για να δούμε τι έχει να μας πει η Κομισιόν. Thank you, Madam. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν συμμερίζεται τον προβληματισμό του εξώτιμου κυρίου Ευρωβουλευτή για την κατάσταση στο Κάμπ Ασραφ. Ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι η κατάσταση εκεί είναι περιπλοκότατη και δύσκολο να εκτιμήσουμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Η Κομισιόν από κοινού με τα κράτη-μέλη είναι παρούσα στο Ιράκ και παρακολουθεί τις εξελίξεις. αλλά δεν έχει πρόσβαση στο Καμπάσραφ που όπως ξέρετε βρίσκεται στα σύνορα με την Περσία. Από τον Ιανουάριο η κυβέρνηση του Ιράκ ανάλαβε πλήρως την ευθύνη για την ασφάλεια στο χώρο αυτό Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι υποχρεώσεις των αρχών να έχουν υψηλό βαθμό προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων του κάθε κρατουμένου. Τον Ιούλιο είχαμε πληροφορίες για το τι έγινε, αλλά από τρίτες πηγές. Δε, σας είπα δεν έχουμε άμεση πρόσβαση. Άρα οι πληροφορίες μας στηρίζονται σε εκθέσεις που παίρνουμε από τον ύπατο αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και από άλλους. Οι εκθέσεις αυτές λένε ότι η προσπάθεια της ε, κυβέρνησης να μπει στο στρατόπεδο οδήγησε σε 11 θανάτους και σε πολλούς τραυματισμούς. Βέβαια μια τέτοια τραγωδία φυσικά απαιτεί επίσημη ανάκριση και η κράτηση ατόμων χωρίς κατηγορία, χωρίς απόδοση κατηγορίας επιμήνης και αυτό είναι απαράδεκτο. Βέβαια το Ιράκ είναι μια επικυρίαρχη χώρα και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να τηρούν, να εξασφαλίζουν μάλλον τάξη σε όλη τη χώρα. Στο Κάμπ Άστραφ, από ό,τι φαίνεται, είναι ένας θύλακας ειδική μορφής μέσα στη χώρα και δεν είναι πραγματικά υπό τον έλεγχο των δημοσίων αρχών. Γι' αυτό το να προωθήσουμε περισσότερο την νόμο και την τάξη για να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη χώρα αυτή η οποία επέφερε τόσο πολλά είναι κάτι το επιβαλόμενο αλλά οι αρχές κατά την άποψή μας είναι υποχρεωμένες να φέρουν σε πέρα στις υποχρεώσεις τους για το πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις διεθνείς συμβάσεις. Η Ένωση θα κάνει ό,τι μπορεί να το τονίζει αυτό στις αρχές και σε υπουργικό επίπεδο και στην τελευταία τρόικα με το Ιράκ στα πλαίσια της συνάντησης Ούγκα το Σεπτέμβριο στις 24 ετέθη το θέμα του στρατοπέδου Άσραφ. Σε άλλο επίπεδο προσφέρουμε βοήθεια στο Ιράκ για εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να εκπαιδευτούν τα διάφορα στελέχη με βάση το πρόγραμμα νόμος και τάξη. Έχουμε πολλές εκδοχές ως προς το τι έγινε στο στρατόπεδο με βάση αυτό που μας είπε η κυβέρνηση, η κίνηση ήταν μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η γη σε βάρος επικυρίαχου εδάφους του Ιράκ. Υπήρξε βία Πάντως εμείς προσπαθήσαμε στις αρχές να περάσουμε το μήνυμά μας ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Παραμένουμε ενεργοί. Επαλαμβάνω το θέμα είναι περιπλοκότατο. Δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς όσον αφορά τα γεγονότα επειδή δεν έχουμε άμεση πρόσβαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κάζακ, υποθέτω, θέλει να κάνει ερώτηση. Да, Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τόσα μας είπε, που μας απάντησε δηλαδή με τόσες λεπτομέρειες. Δίχως άλλο, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα από την αρχή της χρονιάς είναι γεγονότα τα οποία μας ανησυχούν. Διότι πρόκειται για αθώους οι οποίοι τελικά γίνονται θύματα, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται προκειμένου να λυθούν γεωστρατηγικά ζητήματα μεταξύ δύο γειτόνων χωρών. Όμως, αυτό που ιδιαίτερα με ανησυχεί και πραγματικά εξεπλάγινα από τις εικόνες που είδα, σοκαρίστηκα μάλιστα, που δείχνανε τις Ιρακινές δυνάμεις να μπαίνουν στο, στο τόπο και την έλλειψη αντιδράσεων από την άλλη μεριά, από πλευράς των Αμερικανών δηλαδή στρατιωτών, οι οποίοι διασφάλιζαν, ε, προστάτευαν μάλλον ε, το στρατόπεδο αυτό. Νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα λοιπόν πρέπει να αντιδράσει, πρέπει να επιβάλλει μέτρα αυστηρά, διότι παραβιάζονται δικαιώματα. Ευχαριστώ πάντως κυρία Πρόεδρε που φροντίσατε να στείλετε επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Σουηδίας και στον Ήπατο Αρμόδιο, προκειμένου να πάει από τον ΟΙΕ μια ομάδα παρατηρητών εκεί επιτόπου και αν γίνει αυτό, ειλικρινά πιστεύω ότι θα έχουμε ήδη μια πιο αντικειμενική εικόνα για την κατάσταση. Οι Ρακίνες αρχές από την άλλη μεριά ίσως έτσι αναγκαστούν να δράσουν. Πάντως, ο ΙΕ και η Σουηδική Προεδρία είναι εκείνοι που μπορούν να μας στηρίξουν, γιατί εμείς δεν μπορούμε να διαφορούμε για την τύχη αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστούμε. Ε, τόσο εγώ όσο την αντιπρόεδρος ε, συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία αποστέλλοντας και μια σχετική επιστολή προς τον Αρμόδιο των Ηνωμένων Εθνών και πράγματι ε, όπως μόλις τώρα πήγε ο κύριος Κάζα ε, η κατάσταση και χειροτερεύει όλο ένα και περισσότερο. Έχουμε λίγο ακόμα χρόνο στη διάθεσή μα ε, και μπορούμε να θέσουμε άλλε δύο ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η συνήθι πρακτική αυτή, αλλά είναι πολύ σύντομε ερωτήσει, σα μπορούμε να το κάνουμε. Ένα λεπτό ή 30 δευτερόλεπτα. Πρώτος ο κύριος Στίβενσον λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σα ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο και παίρνω το λόγο ως ε, πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας ε, για το Ιράκ και ειδικότερα για αυτό το θέμα θα ήθελα να πω κάτι εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Συζητούμε λοιπόν εδώ το στρατόπεδο Άστραφ στο οποίο ε, έχουμε 3.500 ε, ε, ανθρώπους από την ομάδα του Μουζαχεντίν του Ιράν που είναι ουσιαστικά πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν καμία προστασία σε αυτή τη φάση οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία και λαμβάνουν την υποστήριξη όλης της κοινωνίας από, το, από τον ευρύτερο χώρο και τους οποίους ε, έχουν, ε, έχουν δοθεί εγγυήσει σε ό,τι αφορά την πλήρη τους ε, προστασία από τον Αμερικανικό στρατό, αλλά έχουν και πλήρες καθεστώς προσφύγων. Καθώς δεν έχει υπάρξει κανένας είδους απειλή για την ασφάλεια ή την κυριαρχία του Ιράκ. Θεωρούνται απειλή για το γειτονικό Ιράν, όπου αποτελούν την κύρια αντιπολιτευτική ομάδα. Και είναι λοιπόν το Ιράν εκείνο το οποίο έχει ασκήσει πιέσει στην Ιρακινή κυβέρνηση τους, ώστε να ελέγξει αυτό το στρατόπεδο. Και θεωρώ πως ε, ε, το Ιράν είναι εκείνο το οποίο επιμένει ε, οι 36 αυτοί κρατούμενοι να παραμείνουν φυλακισμένοι και να απελαθούν στο Ιράν, στο οποίο είναι σίγουρο ότι θα βασανιστούν και θα εκτελεστούν. Βασικά αν τα πράγματα γινόταν σύμφωνα με τα όσα επιθυμεί το Ιράν και οι 3.500 φιλοφιλούμενοι στο στρατόπεδο Αστρεφτά ε, απελάβνονταν ε, στο Ιράν προκειμένου να εκφραστούν εκεί. Και βλέπουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία ε, συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια ότι είχαμε ένα μείζον ψήφισμα στο Κοινοβούλιο το οποίο αγνοούν οι και έχουμε τρεις τώρα αποφάσεις από τα δικαστήρια τα οποία ε, των δικαστηρίων ε, του ίδιου του Ιράκ έτσι που ε, προβλέπουν ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν αυτού του 36 κρατούμενοι οι οποίοι είναι, βρίσκονται στην 24η ημέρα της απεργίας πείνας τους με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να κοντεύουν να πεθάνουν και παρόλα αυτά δεν έχουν απελευθερωθεί αλλά πραγματικά θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε έντονα στην Ιρακινή κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στίβενσον. Ε, ως ε, πρόεδρος της σημερινής συνεδρίασης θα πω ε, ε να υπενθυμίσω πως ε, ζήτησα από τους συναδέλφους να είναι σύντομοι. Αντιλαμβάνομαι πως ε, υπάρχουν εδώ έντονα συναισθήματα, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να περάσουμε δηλαδή στο θέμα της Στριλάνκα. Άρα λοιπόν ο κύριος Μοντάντο θα πάρει το λόγο και συνέχεια η κυρία Σύγκλαρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Για να επεκτείνω λίγο το ζήτημα της ε, πρόσβασης. και με βάση τα όσα έχετε παρατηρήσει, ποια θεωρείτε πως θα ήταν η κατάλληλη ε, κατάλληλη δράση ή τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε, ούτως ώστε να μας επιτραπεί η πρόσβαση εκεί. Στο, Ναι, πολύ σύντομη ερώτηση και πολύ αυστοχή. Η κυρία Σίνκλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάζακ που έθεσε αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα. Ε, ενημερώθηκα για αυτές τις ακρότητες οι οποίες έλαβαν χώρα τον Ιούλιο ε, και πραγματικά ήταν ε, πάρα πολύ ανησυχητικά όλα αυτά. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη γιατί όλα τα σχόλια που ήθελα να κάνω έγιναν ήδη από τον συνάδελφο και συμφωνώ μαζί του και επίσης αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Ιράκ είναι κυρίαρχο κράτος και έτσι τα πράγματα είναι δύσκολα για μας αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρατηρούμε και βέβαια προφανώς και να θέτουμε τα ζητήματα αυτά με τον τρόπο στους συναδέλφους μας, στους ομολόγους μας στα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκυλά. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεται για να επιστήσουμε την προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο Άστρα. Η απάντηση μας έδωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητική γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ε, ως δικαιολογία το γεγονός ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη όπως μας είπε. Ε, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου είναι πολύ ε, σαφές. Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για 36 πρόσωπα, 36 άτομα τα οποία για τα οποία έχει, δοθεί, έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Άρα θα πρέπει εδώ να αναλυθεί δράστη εγώ ω ε, μέλος της αντιπροσωπείας ε, για τη σχέση με το Ιράκ είχα επισκεφθεί το στρατόπεδο Άστραφ με, πέρυσι μαζί με τρεις συναδέλφους. Και πρέπει να πω πως είναι ένα υποδειγματικό στρατόπεδο το οποίο προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση του να φέρει μια δημοκρατική αλλαγή στο Ιράκ. Είναι ε, τα άτομα εκείνα τα οποία πρώτα αποκάλυψαν στον κόσμο ε, την ύπαρξη ε, των προσπαθειών για κατασκευή πυρηνική βόμβα από το Ιράν. Οπότε θα πρέπει να του είμαστε ευγνώμονε και να του ευχαριστούμε με κάθε τρόπο. Σα ευχαριστούμε. Ναι. Ε, Προφανώ μπορούμε να κινηθούμε εδώ περαιτέρω και θα ζητήσουμε και από τον πρόεδρο να επανθυμίσει για μία ακόμα φορά αυτό το ζήτημα στην ελληνική πλευρά. Θα ήθελα να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Ναι. Αυτή μια τέτοια κατάσταση, βέβαια, για μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ μια απολύτω ικανοποιητική απάντηση. Αλλά στις 24 Σεπτεμβρίου η Τρόικα από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση έδεσε στο ΙΡΑΚ αυτό το ζήτημα. Ε, ειδικότερα το ζήτημα της απελευθέρωσης των 36 αυτών κρατουμένων. Ίσως πράγματι θα πρέπει να θίξουμε αυτό το ζήτημα και στην Αμερικανική πλευρά, όπως είπε η Αλλά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς ε, πρέπει να βασιζόμαστε στο, στο γραφείο του υπατέρμοστη για τα ανθρώπινα και στα όσα έχει το ICRC. Δεν ε, μεριζόμαστε απολύτω ε, την άποψη ότι πρόκειται για ένα υποδειγματικό στρατόπεδο το οποίο κατευθύνεται ε, προς τον εκδημοκρατισμό και του Ιράν. Μιλάμε για... Μιλάμε για μια οργάνωση η οποία μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζει να υπάρχει στον κατάλογο αυτό ε, της, ε, τον ΗΠΑ αλλά και στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη οργάνωση, θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό και ταυτόχρονα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι δύσκολο για τις Ιρακινές αρχές να παραδεχτούν ότι πράγματι υφίσταται ένα στήλακας μέσα στη δική τους επικράτεια ε, χωρίς όμως να μπορούν να σκίσουν έλεγχο, να βρίσκεται υπό τον έλεγχό του αυτό ο θύλακας. Ε, παρόλα αυτά, ε, οι αρχέ αρχές θα πρέπει να σεβαστούν πλήρως τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα στον ανθρωπιστικό χώρο. Αλλά η κατάσταση είναι δύσκολο να αξιολογηθεί λεπτομερώς και εμείς συνεχίζουμε να φύγουμε αυτό το ζήτημα στους Ιρακινούς και θα θέλαμε να βεβαιώσουμε τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου ότι δεν ξεχνούμε, δεν προσπερνούμε την πραγματικά τραγική κατάσταση που επικρατεί αυτό το στρατόπεδο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τιμάντζη για αυτέ τι απαντήσει που έδωσε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις πρόσθετες πληροφορίες. Προφανώ υπάρχουν διστάμενε απόψει σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα αλλά όπως είπα είναι απαραίτητο να ε, γίνει σεβαστό το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο την τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, εδώ ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε σήμερα εδώ για να σε ενημερώσει ε, σε σχέση με τα όσα πράττει. Ε, περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διαταξής μας που είναι μια δημόσια ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Στρι Λάνκα. Έχουμε μαζί μας τέσσερις ομιλητές ο πρώτος ομιλητής είναι ένας εμπειρογνώμονας ε, μετά έχουμε τον διευθυντή της αρμόδιας μονάδας της International Crisis Group. Μετά έχουμε μια κατάθεση, αν θέλετε, εδώ από τον Σουνάντα Ντεσάπρια, έναν δημοσιογράφο και ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα από αυτή τη χώρα. Θα λάβουμε επίση την διεθνή πτυχή του ζητήματο από τον Αντουάν από τον συντονιστή για τις ανθρωπιστικές δράσεις ε, των Ηνωμένων που εντρεύει εδώ στις Βρυξέλλες και μετά θα ακούσουμε και τον David Tier ως πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας ε, μιλήσει σε σχέση με το GSP Plus και τις ε, ε, τελωνιακές συμφωνίες που έχουν χώρα και επίσης θα ακούσουμε και δύο λόγια από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Τριλάνκα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους βασικούς ομιλητές να περιοριστούν σε 10 λεπτά σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις τους ε, για να έχουμε και κάποιο χρόνο να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να δώσω λοιπόν καταρχήν τον λόγο στον Άντρου Στρόλαν από την International Crisis Group. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τέσσερις μήνες τώρα. Έχει λήξει ο εμφύλιος πόλεμος στην Σρι Λάγκα. Από τότε 250.000 Σταμούλ έχουν φυλακιστεί, είναι σε στραδόπεδα, στη, στο βόρειο κομμάτι της χώρας. Τους έχει περιορίσει το κράτος με σύρματα γύρω-γύρω και είναι έτοιμοι να πυροβολήσουν κάθε έναν που προσπαθεί να αποδράσει από εκεί. Περιορίζεται λοιπόν η ελευθερία τους, παραβιάζονται οι νόμοι, τόσο οι εθνικοί όσο και οι διεθνείς. Η κατάσταση βέβαια χειροτερεύει συνέχεια, οι ιατρικές υπηρεσίες δεν είναι αρκετές, η γενή δεν είναι καλή, ε, αυξάνεται ο πληθυσμός συνεχώς κλπ. κλπ. Οι στρατιωτικοί εμποδίζουν ε, τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, όσο και τον ΟΗΕ, την υπεύθυνη υπηρεσία για τους πρόσφυγες, να παρέμβουν. Η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλές υποσχέσεις τους τελευταίους τέσσερις μήνες για το πώς, πότε οι μετατοπισμένοι αυτοί θα φεθούν ελεύθεροι. Είπαν σε έξι μήνες, μετά είπα στο τέλος της χρονιάς, μετά είπα τον Ιανουάριο, αλλά τίποτα. Πριν από τρεις εβδομάδες, ναι, πριν από τρεις εβδομάδες, το Κολόμπο είπε ότι η κυβέρνηση θα ελευθέρωνε 10.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Δεν έγινε αυτό όμως. Ανακοίνωσαν ότι άφησαν 10.000, αλλά τελικά τι έκαναν, τους μετέφεραν από έναν καταβλισμό σε έναν άλλον. Άρα η αξιοπιστία των υποσχέσεων αυτών είναι προφανές ότι δεν υπάρχει δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτά που μας λένε. Στο τέλος του πολέμου είχαμε ακούσει διάφορα νούμερα από τον ΟΗΕ. 289 ήταν μετατοπισμένοι εσωτερικά από τον πόλεμο. 10.000 από αυτούς, 289.000 προφανώς, ε, φαινόταν ότι είχαν ε, σχέσεις με τους ε, τρομοκράτες επαναστάτες και είχαν κρατηθεί με την κατηγορία ότι είχαν τέτοιες σχέσεις με τρομοκράτες. Ε, άλλοι τόσοι μπόρεσαν να φύγουν, είχαν χρήματα, είχαν γνωστούς, συνδέσεις κτλ. στο καλύτερο για αυτούς και 6.000 είχαν κατασταθεί αλλού. Τα καλύτερα νούμερα που έχουμε, αλλά βέβαια δεν συμπίπτουν πάντα τα νούμερα. Πολλές φορές βασιζόμαστε στα νούμερα που δίνει η κυβέρνηση. 264.000 όμως σήμερα. Οι περισσότεροι από αυτούς αθώοι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τα σπίτια τους, βρίσκονται σε καταβλισμούς και δεν μπορούν να φύγουν. Ακόμα και είπα ότι η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δεν έχει μπορέσει να κάνει τίποτα. Ζητάνε να πάνε, αλλά ποτέ ποτέ δεν τους δόθηκε η άδεια να πάνε και να επισκεφθούν τους καταβλισμούς αυτούς, ούτε καν τους 10.000 που κρατούνται, επειδή ε, τους κατηγορεί η κυβέρνηση ότι έχουν σχέσεις με τρομοκράτες. Έπειτα, τι λένε, λένε, πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να εξοδετερωθούν οι νάρκες, αλλά μπουρδες, διότι θα μπορούσαν να πάνε σε συγγενείς τους, θα μπορούσαν να πάνε σε φίλους τους που ζουν κανονικές ζωές σε χωριά, σε πόλεις, στην Σρι Λάγκα και που εκεί δεν έχει νάρκες. Ε, η δεύτερη αιτία, που, η δεύτερη δικαιολογία που δίνει είναι ότι για τους 264.000 πρέπει να ελέγξουν πρώτα μήπως έχουν σχέσεις με τους τρομοκράτες. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει κανένα νούμερο, κανένα στοιχείο για κανέναν, για πόσους έχει ελέγξει ήδη και η πατερμοστή του ΟΗΕ δεν έχει μπορέσει να ελέγξει τίποτα από όλα αυτά. Και όταν μιλήσαμε στου καταπλησμού με του ανθρώπου, οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα ότι γίνεται αυτό, ότι δηλαδή κάποιο ελέγχει τι διασυνδέσει του. Και στο κάτω-κάτω τέσσερι μήνε έχουν περάσει. Αν τέσσερι μήνε κάνει αυτό τον έλεγχο κυβέρνηση, ε, τέλο πάντων κάποιοι δεν θα έπρεπε να είχαν ελευθερωθεί από αυτού. Οι πρόσφατε υποσχέσει έτσι και αλλιώς αφορούν ε, μερικούς μικρούς καταβλισμούς, όχι τις ε, μεγάλες αυτές ε, τις μεγάλες συγκεντρώσεις αυτές πληθυσμού. Ε, λένε δηλαδή ότι μπορούν να τους δίνουν κάποια πά για μια μέρα. Ναι, αλλά αν μπορούν για μια μέρα να καταλήψουν του καταβλισμού και να κινηθούν ελεύθερα, γιατί να μην μπορούν συνέχεια να το κάνουν. Πάντω, ούτε υποσχέσει τη κυβέρνηση, ούτε για απελευθέρωση, ούτε για βελτίωση, ούτε τίποτα, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Και η αρμόδια του Ιωτε δηλαδή για την μετατόπιση πληθυσμού, ένα ανακοινωθέν. Ε, ξέρετε, φαντάζομαι ο συνάδελφο εδώ θα σας μιλήσει γι' αυτό. Και λέει εκεί, και τώρα τον παραθέτω, ότι είναι απαραίτητο αμέσως να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ε, λιγοστέψει ο κόσμος που κρατείται στου καταβλισμούς αυτούς, να ελευθερωθούν οι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει σε θελοντική βάση να μπορούν και ελεύθερα να φύγουν με ασφάλεια να φτάσουν στα σπίτια τους. Και πρέπει να τους δοθεί ευκαιρία να ζήσουν όπως θέλουν με συγγενείς τους, με δικούς τους, ελεύθερα. Να ανοίξουν οι πύλες, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν χωρίς να κινδυνεύουν να φάνε ένα βόλι στην πλάτη φεύγοντας. Έχουμε ακούσει και πολλά σχόλια για την πικρία στους Ταμούλ. Βλέπετε, είναι μία κρίση που δεν είναι μόνο ανθρωπιστική, ο πρόεδρος των ΗΕ ακριβώς σε αυτό αναφέρθηκε. Είπε ότι κρατώντας πάνω από 25.000 ανθρώπους εκεί, χωρίς ε, κατηγορία, είναι, δημιουργεί μια τέτοια δυσαρέσκεια που θα οδηγήσει στην επόμενη εθνική σύραξη στη Σρι Λάγκα. Και αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Όσο περισσότερο κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι, χωρί κατηγορία, μέσα στου καταβλισμού αυτού, καταλαβαίνετε πόσο πιο πολύ απογοητεύονται, θυμώνουν ενοχλούνται και καταλαβαίνετε αυτό κινδυνεύει να οδηγήσει σε ένα νέο εμφύλιο πόλεμο εκεί. Και αυτό λέμε εδώ και χρόνια. Ελπίζουμε τώρα που έχουμε το μήνυμα και από τον ίδιο τον ΟΗΕ να το προσέξει η διεθνή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και τα κράτη-μέλη τι μπορούν να κάνουν. Είναι περιορισμένη η επιρροή που μπορούν να έχουν στην κυβέρνηση άλλοι θα μιλήσουν για το GSP συν. Κοιτάξτε, το βασικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με καθαρό λόγο και να ζητήσει την ελευθερία διακίνησης αμέσως. Αυτό. Δεύτερον, να ζητήσει πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ανθρωπιστικών οργανώσεων επιτόπου, να μπορούν να πάνε, γιατί επίτηδες μας κρύβει πληροφορίες η κυβέρνηση. Τρίτον, αφοπλισμός ε, προγράμματα αποκατάστασης να γίνουν μόνο με τη συμμετοχή του ΟΗΕ, της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Προς το παρόν υπάρχει χρηματοδότηση για κάποια προγράμματα, αλλά δεν συμμετέχει ο ΟΗΕ. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα νομικό πλαίσιο. Και αυτό είναι αρνητικό. Γι' αυτό θέλουμε ό,τι προγράμματα λαμβάνουν χώρα να έχουν και τη συμμετοχή του ΟΗΕ. Τέσσερα να πιέσουμε για χρονοδιάγραμμα. Να μην αφήσουμε τα στρατόπεδα αυτά, τους καταβλισμούς αυτούς, να παραμείνουν και να γίνουν κάτι μόνιμο, μια μόνιμη δοή. Τέλος, υπάρχει και μια άλλη τραγωδία και εδώ όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να μπορούν να επηρεάσουν ώστε η κυβέρνηση να κάνει πραγματικότητα τις υποσχέσεις της. Είτε από τον Ιούλιο είπε στο Διεθνές Μεθοδικό Ταμείο 78% των ε, εσωτερικά μετατοπισμένων θα τους ελευθερώσει σε τέσσερις μήνες. Αλλά η διαδικασία αυτή δεν έχει καν ξεκινήσει οι δωρητές δεν θα πρέπει να δώσουν τίποτα αν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο με διαβουλεύσεις ε, με όλη τη χώρα. Τα χρήματα που δίνονται από διεθνείς δωρητές δεν πρέπει να αποσταθεροποιήσουν περισσότερο την κατάσταση. Γιατί σας είπα, ετοιμαζόμαστε για τον νέο φίλιο πόλεμο, έτσι όπως πάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. κύριε Στρελάνη για τις πρακτικές αυτές τις προτάσεις σας. Φυσικά αυτή η κατάσταση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις, στη μακρόπνοη προοπτική για ειρήνη. Ο κύριος Ντεσάπριο, δημοσιογράφος και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας δίνουμε 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, είμαι δημοσιογράφος, είμαι από το Σρι Λάγκα και είμαι αυτοεξόριστος εδώ και έξι μήνες στην Ευρώπη επειδή απειλείται η ζωή τους πολύ επειδή απειλείται η ζωή πολλών δημοσιογράφων και ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λάγκα όπως και η δική μου. Θα προσπαθήσω να, θα προσπαθήσω να αναφερθώ στην καταστολή στο Σρι Λάγκα, τι έγινε μετά το πέρας του πολέμου το Μάιο και ποιες είναι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές που μπορεί να προτείνει η Ένωση στη Σρι Λάγκα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο πόλεμος κράτησε περίπου 30 χρόνια. Οι ένοπλες δυνάμεις και ο στρατό τη χώρα έχουν όλη ευθύνη για δολοφονίε δημοσιογράφων. Όχι μόνο οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, αλλά όλε οι ένοπλε ομάδε Συμπροβαίνουν και τους ε, τον Πλευθερικό Στρατό του Ταμίλ. Είναι όλοι συνυπεύθυνοι για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε αποδείξεις για εκατοντάδες δολοφονίες τα τελευταία 30 χρόνια. Από τις δολοφονίες αυτές 34 είναι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν από τον Απρίλιο του 2004 που έχουμε την κυβέρνηση αυτό 34 δημοσιογράφοι δολοφόνηκαν δεκάδες έχουν απαχθεί δεκάδες βρίσκονται στις φυλακές και εκατοντάδες απειλούνται τους απειλούν θα τους σκοτώσουν Εβδομήντα δημοσιογράφοι τα τελευταία τρία χρόνια έφυγαν από τη χώρα. Οι περισσότεροι, οι περισσότεροι από αυτού ζουν στην Ευρώπη. Όλοι όταν τελείωσε ο πόλεμο τέλο Μαΐου θεωρήσαμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση Όμω, αν δείτε τι συνέβη στους 4-5 μήνε, πέντε δημοσιογράφοι έχουν απαχθεί ο ένα τραυματίστηκε σοβαρά και ένα πάρα πολύ γνωστό δημοσιογράφος πριν από δύο μέρε, μια γυναίκα δημοσιογράφος που οργάνωσε μια διαμαρτυρία λόγω τη καταστολή στα μέσα ενημέρωση στην Ισλάκα, απειλήθηκε με απαγωγή. Πήγαν στο σπίτι της και της το είπανε. Το γράψαν αυτό οι εφημερίδες χθε. Από τις 34 αυτές δολοφονίες ούτε μία δεν αποτέλεσε αντικείμενο ανοιχτής ανάκρισης. Ούτε μία έκθεση. Ούτε ένα δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με αυτό. Δεν κατα... καταδικάζω την κυβέρνηση για τις δολοφονίες, αλλά είναι ευθύνη της κυβέρνησης να κάνει ανάκριση για τις δολοφονίες αυτές. Κανένα δεν μπορεί να πει ότι λόγω του πολέμου δεν μπορούν να γίνουν ανακρίσεις. Η κυβέρνηση, ο πρώην Πρωθυπουργός, συγγνώμη, πρώην Εξωτερικών, έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλοί πρώην πρόσωπο εξωτερικών, αρχηγός του στρατού κλπ. Η κυβέρνηση βρήκε ποιοι έκαναν αυτές τις δολοφονίες. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση μπορεί να βρει ποιο είναι υπεύθυνο για αυτέ τι δολοφονίε και αυτοκτονίε όπω χαρακτηρίστηκαν μερικέ, γιατί δεν μπορεί να βρει ούτε έναν ένοχο για τις δεκάδες δολοφονίες δημοσιογράφων. Αυτό λέμε στην κυβέρνηση. Συντήσουμε τον πρόεδρο, πολιτικούς της κυβέρνησης και λέμε τουλάχιστον ας ανακριθεί, ας γίνει ανάκριση για μία περίπτωση έτσι ώστε να φανεί ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται υπέρ του κράτους δικαίου. Δυστυχώς αυτό ακόμα δεν έχει συμβεί. Ατιμορρησία λοιπόν στο Σρι Λάγκα Τι λέει η κυβέρνηση. Ο υπουργό τύπου είπε τα εξή. καμία τηλεόραση δεν καταδίκασε τι ελληνές επιθέσεις στην Παλαιστίνη. Όλος ο κόσμος το καταδίκασε. Και καλό τα μέσα ενημέρωσης να είναι προσεκτική όταν μιλάνε για θέματα που είναι επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια. Και ένας άλλος υπουργό είπε τα μέσα ενημέρωσης Μερικοί δημοσιογράφοι είναι προδότες και πρέπει να συντρίψουμε αυτά τα καθήκια. Κυριολεκτικά αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε ο υπουργό μιλώντα για δημοσιογράφους. Και ο αδελφός του Πρόεδρου ε, Υπουργό Άμυνα είπε στην τηλεόραση ανοιχτά. Εγώ αναγνωρίζω δύο κατηγορίες ανθρώπων. Προδότες και αυτοί που καταπολούν πολεμάνε την τρομοκρατία. Έτσι βλέπουν λοιπόν η κυβέρνηση τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρω... Η κυβέρνηση δηλαδή δεν δέχεται ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Οι Ταμίλοι είπαν ότι είχαν 400.000 άτομα στο στρατό τους. Η κυβέρνηση είπε ότι έχουν μόνο 10.000. Τελικά ήταν 300.000. Επειδή δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι παρατηρητές, δεν ήταν δυνατόν όλα τα άτομα αυτά να βρούνε στέγη όταν το χρειάστηκαν. Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι απολύτως αναγκαία σε κάθε χώρα για την ενημέρωση, σε οποιαδήποτε χώρα όπου υπάρχει κράτος νόμου και δικαίου. Η Ένωση πρέπει να ανησυχεί για την κατάσταση στο Σρι Λάνκα. Πρόσφατα ένας δημοσιογράφος Ταμίλ δικάστηκε σε καταναγκαστικά έργα 20 χρόνια και ένα από την κυβέρνηση είπε στην Αλτζαζίρα ότι έγραψε άρθρα κατά της κυβέρνησης και έπρεπε να φυλακιστεί. 20 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Επειδή έγραψε δύο μόνο άρθρα. Ενώ άλλοι από το ίδιο στρατόπεδο πλήρωσαν 20.000 ρούπιε, δηλαδή τίποτα, και έχουν βγει από τη φυλακή ή έχουν γίνει και υπουργοί. Και ο άλλο έγραψε δύο άρθρα και έφαγε 20 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Ζητούμε από την κυβέρνηση να απελευθερωθεί αυτό ο δημοσιογράφο. Πρέπει να κάνουμε καμπάνια να απελευθερωθεί. Σα μοίρασα το κείμενο με, τις με τα βραχυπρόθεσμα αιτήματά μα. Να σταματήσει οποιαδήποτε απαγωγή, όχληση, άσκηση πίεση και βία σε βάρο των μέσων ενημέρωση εκ μέρου όλων των μερών στη χώρα. Μια διαφάνεια και έγκαιρη ανάκριση για τι δολοφονίε δημοσιογράφων και των οικογενειών του. έτσι ώστε να ενισχυθεί η ελευθεροτυπία και η ελευθερία έκφρασης και να καταργηθεί η λογοκρισία. Μακροπρόθεσμα, κύριε Πρόεδρε του Ευρωκοινοβουλίου, κατά επανάληψη έκανε συστάσει στην κυβέρνηση με, με αποστολή παρατηρητών για τις εκλογές τα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης να γίνουν εξάρτητα. Αν θέλετε να έχουμε αλλαγές στην συμπεριφορά του μέσα ενημέρωσης πρέπει να αλλάξει αυτός ο, ο ελεγχόμενος τύπος σε ελεύθερο τύπο. Μακροπρόθεσμα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης. Το προβλέπει το Σύνταγμα. Αλλά αυτά που γίνονται δεν συμφωνούν με τις διεθνείς πρακτικές. Βράχει πρόθεσμα, θέλουμε να δείτε τα μέτρα που σας ανάφερα πριν και τα μακροπρόθεσμα, να έχουμε ελευθερία και δημοκρατία στη Σρι Λάγκα. Και τελειώνω με ένα λεπτό για τα στρατόπεδα IDP, πρόσβαση στα στρατόπεδα. Όσοι ευρωβουλευτές, θα σας παραξενέψει αυτό που θα σας πω, η κυβέρνηση οι σύζυγοι τους, τα παιδιά τους μπορούν να πάνε στα στρατόπεδα, αλλά ούτε ο επικεφαλής αντιπολίτευσης δεν επιτρέπεται να μπει. Και βουλευτές που εκπροσωπούν αυτούς τους ανθρώπους, τα Μίλ και άλλους, βουλευτές, επαναλαμβάνω, δεν τους επιτρέπεται μέχρι τώρα να μπουν στα στρατόπεδα, ούτε ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος δεν επιτράπει να μπει τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Ενώ οι πολιτικοί, οι γυναίκες, τα παιδιά τους πάνε και μοιράζουν διάφορα πράγματα και στα στρατόπεδα τη κυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση, να ξέρουμε τι έγινε και στη διάρκεια του πολέμου, τι έγινε με τους ανθρώπους αυτούς. Χωρίς ελεύθερο τύπο, χωρί πρόσβαση στα στρατόπεδα δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, Σα ευχαριστούμε και εμείς κύριε Ντεσάπιαρ. και για το γεγονός ότι μας αναφέρατε τόσο κάποιους ε, βραχυπρόθεσμος όσο και κάποιους μακροπρόθεσμος ε, στόχους. Θα πρέπει πράγματι να ε, επιδείξουμε προσοχή προκειμένου να επιτευχθούν. Και βέβαια τα αιτήματά σας μας επενθυμίζουν τα όσα αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους που είχαμε χθες εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, όπου ήταν παρόμοια αυτά που ακούγαμε, ότι δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση τη νόμη και ούτω καθεξή. Τώρα θα ακούσουμε λοιπόν την άποψη ε, από το γραφείο του συντονιστού ε, για την ανθρωπιστική δράση από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, κύριο Σαρατουάν, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σα ε, ευχαριστώ που αναφέρεστε στα ανθρώπινα δικαιώματα και διοργανώνετε αυτή τη συζήτηση. Σήμερα δεν θα ήθελα να προβώ σε περιγραφή της κατάστασης ε, καθώς ε, το έπραξαν ήδη οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Απλά θα ήθελα να αναφερθώ στο τι κάνουμε εμείς από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, την εξέδωση κατοικιών. Ε, ακούσαμε τα κύρια ζητήματα σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στους καταβλισμούς ε, και πώ μπορεί να επιληθεί η κατάσταση. Όπως ακούσατε, ε, ε, υπάρχουν υπερβολικά πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτούς τους καταβλισμούς ειδικά όταν αυτοί βρίσκονται σε, είναι περιφερειακοί και σε αυτές τις περιπτώσεις ε, δεν μιλάμε απλώς ε, για τον περιορισμό των δικαιωμάτων μετακίνησης αυτών των ατόμων αλλά το γεγονός ότι έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς τους καταβλισμούς όλα αυτά τα άτομα ενώ ταυτόχρονα πλησιάζει η εποχή των μουσώνων δηλαδή των δυνατών βροχών ε, με κάποιες πρώτε ενδείξει που δείχνουν ότι καταστράφηκαν κάποια τμήματα αυτών των καταβλισμών ένα γεγονό το οποίο ε, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση αυτών των ατόμων. Ε, είναι λοιπόν πολύ δύσκολες οι συνθήκες και μας ανησυχεί πολύ η φύση αυτών των καταβλισμών ε, όπως ε, ανέφερε ο συνάδελφο από την International Crisis Group και ο δημοσιογράφος από τη Σρι έχουν ε, ασκηθεί πολύ μεγάλε πιέσει από τη δική μα ε, πλευρά στην κυβέρνηση τη Σρι γιατί είμαστε πολύ απογοητευμένοι σε ό,τι αφορά την πρόοδο ή τη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση αυτών των ατόμων, καθώ δεν δεν έχουν το δικαίωμα μετακίνησης εκτός από κάποιες ειδικές ομάδες όπως η ΕΡΙΣ χαιρετίζουμε την απόφαση που έλαβε ο Πρόεδρος ε, του να έχουν το δικαίωμα τα άτομα αυτά να ε, εγκαταλείψουν του καταπληκτισμού τη οικογένειά του, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά την εφαρμογή αυτή τη πολιτική. Ακούσαμε και ακόμα ακούμε. Ε, δηλώσαμε επανειλημμένα προς την κυβέρνηση της Λάγκα να σεβαστεί και τα δικαιώματα αυτών των ε, ατόμων και μάλιστα πριν καν από την επιστροφή τους ε, στις ε, κατοικίες τους. Το Ηνωμένα Έθνη έχουν διάφορους τρόπους να ασκούν τις πιέσεις τους και όπως γνωρίζετε ο γραμματέας σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αποθέσεις, ο Λίν Πάσκο, επισκέφθηκε τη Σελάνκα περίοδο 16 έως 19 Σεπτεμβρίου και ενημέρωσε το Walt Kelling, τον εκπρόσωπο δηλαδή του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος και εκείνος επισκέφθηκε τη Στριλάνκα Και έχω εδώ ε, ε, μπροστά μου την ανακοίνωση ε, τύπου ε, ότι πριν από δύο ημέρες όπου αναφέρεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο το τι ακριβώς ζητάμε. Στη Νέα Υόρκη τώρα ο Γενικός Γραμματέας ε, συναντήθηκε με τον Υπουργό της Στριλάνκα και ε, συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να παρακολουθούμε διεθνώς την κατάσταση του ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι οι IDP, τα άτομα δηλαδή αυτά, θα επιστρέψουν στις κατοικίες τους ε, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα. Γιατί δεν μας ε, ανησυχεί μόνο η τωρινή κατάσταση, μα ανησυχεί και η μελλοντική κατάσταση. Ε, η κυβέρνηση της Σιλάνκα είχε δεσμευτεί να επιστραφεί ή να επιτρέψει να επιστρέψουν το 70% των ΑΕΤΠΙΣ στις κατοικίες του στο Βορρά, όμως η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα κοινοποιήσει ένα πλήρες σχέδιο επιστροφής ε, αυτών των ατόμων στις κατοικίες τους, πράγμα που καθιστά το δικό μας σχεδιασμό και τη δική μας υποστήριξη απέναντι στην κυβέρνηση της ιδιαίτερα δύσκολο. Οπότε την καλούμε την κυβέρνηση τη Σρι γιατί αυτό το κάναμε, δηλαδή αυτή την έκκληση την απευθύναμε και σε διάφορε συναντήσει μα να ε, κοινοποιήσει στην διεθνή κοινή γνώμη αυτό το σχέδιο επιστροφή και να συμβουλευτεί και τι διάφορε ανθρωπιστικέ ε, οργανώσει, οι οποίε είναι παρούσες αυτή τη στιγμή στη Σρι Αναμένουμε να δούμε μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Σρι Λάγκα και Ευρωπαϊκή Ένωση και των ανθρωπιστικών οργανώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ενό ε, στενού διαλόγου σε ό,τι αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να δοθεί πρόσβαση σε όλες τις ε, περιοχές όπου είχαν λάβει χώρα οι μάχες ε, και θα πρέπει να δοθεί και πρόσβαση στα μέσα και σε αυτούς τους καταβλισμούς ώστε να ε, ε, συλλεγούν κάποιες καταθέσεις και να διασφαλιστεί η προστασία αυτών των ατόμων. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής αυτής και αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που κάνει το Κοινοβούλιο ε, για να διασφαλιστεί ανθρωπιστική βοήθεια προς ε, αυτούς τους ε, ανθρώπους, ειδικότερα η ΕΚΟ, δηλαδή η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει παράσχει εξαιρετικό έργο. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε την εθνική συμφιλίωση και την ειρήνη στη Στριλάνκα, για την οποία είναι απαραίτητη η σωστή μεταχείριση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και επισοφή των IDP των ε, εμένοντων δηλαδή σε αυτού του ε, καταβλισμού και θα πρέπει να σημειωθεί ταχύτερη πρόοδο σε ό,τι αφορά την ελευθερία μετακίνησή του και την επιστροφή του. καθώς ε, αν δεν γίνει αυτό δεν θα είναι εύκολο να συνεχιστεί η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι απαραίτητο οι δωρητές όσο και τα κύρια κράτη που εμπλέκονται εδώ, δηλαδή και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο να παρακολουθούν τα όσα πράττει η κυβέρνηση της ε, Στριλάνκα αλλά και να το κάνει ε, να, ό,τι πρέπει να το πράττει σύμφωνα με το Διεθνέ Ανθρωπιστικό Δίκαιο σε αυτό το τομέα και την εθνική τη νομοθεσία και σπουσόμαστε και δική μα ε, βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτήν την κύριε Ζεράρ για αυτήν την παρουσίαση η οποία ασχολήθηκε με κάποιους από τους δυνατούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρασχούμε βοήθεια να αξιώσουμε πράγματα από την ε, Στριλάνκα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές ε, τη χάνουν βασμό σε αυτή τη χώρα. Η τέταρτη παρουσίαση που θα ακούσουμε είναι αυτή από το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ε, μπορεί να μας πει περισσότερα σε ό,τι αφορά το σύστημα GSP+, δηλαδή τις θελονιακές συμφωνίες. Κύριε Στέλφ και ο κύριο ε, Τίμα θα μιλήσουν εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινάμε όμω με τον κύριο Τίμαν. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μας απασχολεί βεβαίως το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο νησί αλλά νομίζω ότι πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανθρωπιστική βοήθεια ιδιαίτερα ε, των ανθρώπων που βρίσκονται κλεισμένοι στους καταβλισμούς. Όπως είπε και συνάδελφος από τα Ηνωμένα Έθνη, σίγουρα είναι με διαφορά το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε. Και ο γενικό Γραμματέα το έχει πει πολλέ φορέ ότι σε διεθνέ επίπεδο είναι μια μεγάλη ανησυχία και υπάρχει και φόβος και ρωτήσαμε σχετικά και του συναδέρφους από το Σρι Λάνκα για το ότι ίσα θα μείνουν στους καταβλισμούς οι άνθρωποι αυτοί. Είτε εκεί που βρίσκονται τώρα ή αλλού. Πραγματικά είναι δυσανάλογο το νούμερο, δηλαδή των ανθρώπων που βρίσκονται στους καταβλισμούς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γενικότερα μιλώντας πάντως, όπως σας είπα, το θέμα το, ανθρωπιστικό μας απασχολεί και έχουμε κάνει πολλές δηλώσεις από αυτού. Ίσως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα είναι ότι ακριβώς δεν είδαμε τίποτα που να ανακουφίζει κάπως τις ανησυχίες μας όσον αφορά το κλίμα τιμωρησίας που επικρατεί. Όντως, το σύστημα τιμωρησίας είναι αυτό που επικρατεί τελικά. Αν η κυβέρνηση σοβαρά θέλει να βοηθήσει τους Ταμούλ, τότε θα πρέπει να μην τους έχει σαν στόχο. Γι' αυτό και λέω ότι η ανθρωπιστική κατάσταση είναι κρίσιμη όχι μόνο τώρα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Αν ε, μειωθούν ε, τα επίπεδα ε, πώς να το πω, παρέτηση των ανθρώπων εκεί, αυτό θα βοηθούσε. Μην ξεχνάμε και 31 Αυγούστου καταδικάστηκε ε, δημοσιογράφος σε 20 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Γιατί, επειδή έγραψε μερικά άρθρα το 2006. Είναι μια φοβερή περίπτωση αυτή. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για την κυβέρνηση και τον δημοσιογράφο, αλλά είναι κάτι που δείχνει τις προθέσεις της κυβέρνησης πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι να κάτσει και να κρίνει και να καταγγέλει την Στριλάνκα. Εμείς θέλουμε να δούμε κάποιο αποτέλεσμα για τους πρόσφυγες και όσον αφορά το κλίμα τιμωρησίας που επικρατεί εκεί. Και το οποίο βέβαια ενδυναμώνεται από τις ρυθμίσεις που περνούν στο νησί. Το κράτος δικαίου θα πρέπει να ισχύσει και αυτό μπορεί να γίνει να αλλάξει το Σύνταγμα με τροπολογίες. Πάνω σε αυτό θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους. Θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσει η κυβέρνηση της Σριλάνκα, ότι δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όλα τα κράτη-μέλη, ότι είμαστε όλοι σοβαροί, ότι θέλουμε μια αντίδραση από την πλευρά τους, γιατί πολλές φορές είχαμε διάλογο στη Σριλανκά, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι ακόμα πρέπει να τους πείσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και οι βελτιώσεις θα γίνουν μόνο αν υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα στα προβλήματα που εντοπίζει η διεθνής κοινότητα. Τώρα, με ρωτήσατε για το σύστημα γενικημένων προτιμήσεων SIN, GSP+. Είναι ένα περίπλοκο σύστημα πράγματι. Είναι μια συμφωνία ουσιαστικά ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένε υποανάπτυξη χώρε. Με επιπλέον υποχωρήσει εμπορικέ πέρα και από το GSP SIN εφαρμόζοντας 27 διεθνείς συμβάσεις. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μία έρευνα όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή τριών από αυτές τις συμβάσεις. Και είναι λυπηρό για μας ότι η Σρι Λάγκα, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε τις προϋποθέσεις του GSP, Plus δεν δέχτηκε να συνεργαστεί στην έρευνα αυτή, ούτε να δεχτεί τους εμπειρογνώμονες ε, με τους οποίους εμείς είχαμε συμβληθεί για να πάνε να κάνουν την έρευνα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν τα αποτελέσματα και τελική απόφαση στην οποία θα καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασιστεί στα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Με την απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που μας φτάνουν από τη Σρι Λάγκα μέσω άλλων διόδων. Όσον αφορά την ίδια την έρευνα, θα ολοκληρωθεί ένα χρόνο μετά το ξεκίνημά της. Αυτή είναι και η νομική απέτηση, δηλαδή μέσα Οκτωβρίου. Ο τύπος ήδη έχει αναφερθεί κάπως σε μερικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση που θα δημοσιευθεί, αλλά τα τελικά μας συμπεράσματα θα δοθούν στο τέλος της έρευνας και ανάλογα με τις αντιδράσεις της Σρι Εμείς θέλουμε να δώσουμε στη Σρι την ευκαιρία να σχολιάσει την έκθεση αυτή. Αν τελικά αποφασίσει η Επιτροπή ότι πρέπει να διακοπεί η συμφωνία αυτή θα το προτείνουμε στο Συμβούλιο Υπουργών και εκείνοι θα αποφασίσουν αν ναι ή όχι θα πάυσουν προσωρινά την συμφωνία αυτή. GSP+. Αν αποφασίσει πως ναι το Συμβούλιο, τότε θα αρχίσει να ισχύει η απόφαση 6 μήνες μετά την υιοθέτησή της. Θέλω εδώ να τονίσω ότι το μέσο αυτό GSP Plus δεν είναι για να τιμωρήσει κανέναν. Όχι, το, θα το κάνουμε σαν κίνητρο για να αλλάξει η κατάσταση εκεί. Αν δεν πάρει μέτρα να αλλάξει την κατάσταση στη Σριλάνκα και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια νέα πρόταση. Κατά τη γνώμη μου, επειδή ακριβώ συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της ε, Σρι θα πρέπει να έχουμε και έναν χάρτη πορείας που θα βοηθήσει και καλύτερες σχέσεις μεταξύ μας. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Ζαντεπάκτ όρισε μια υπουργική ομάδα όσον αφορά την έρευνα αυτή για το GSP και από ό,τι καταλαβαίνουμε στόχος της είναι να δώσει μια απάντηση στην έκθεση που ετοιμάζουν οι πυρογνώμονές μας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η αντίδραση αυτή βέβαια έρχεται κάπως αργά, γιατί μόνο δύο εβδομάδες μένουν. Μπορώ όμως να υπογραμμίσω ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για άλλη μια φορά είναι συγκεκριμένη πρόοδο. Και αυτή η πρόοδος θα πρέπει να δείχνει ότι η Σρι Λάγκα έχει αναλάβει τα βήματα τα οποία πρέπει για να συμμορφωθεί με τον κανονισμό και τις ρυθμίσεις του συστήματος γενικών προτιμήσεων. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ίσως Πριν ακούσαμε τον, τον κύριο Τίμας να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της πρεσβείας της Σρι που επίσης θα έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του, όπως και άλλοι μας προσκεκλημένοι. Καλώς ήρθατε. Θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες από τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από πλευράς μας, έτσι δεν είναι. Παρακαλώ. θα μου επιτρέψετε καλύτερα να ακούσω τα πάντα και να απαντήσω μετά μια και καλή, γιατί όντω υπάρχουν πολλά ζητήματα και θα ήθελα να μπορέσω να απαντήσω σε όλα στο τέλος. Και καταλαβαίνετε ότι αφού πρέπει να απαντήσω σε μια μισή ώρα περίπου συζήτηση για τέσσερα τουλάχιστον μεγάλα θέματα, όπως σας ζήτησα και πριν, παρακαλώ δώστε μου λίγο παραπάνω χρόνο για να είναι δίκαιο να μπορέσω να απαντήσω σε όλα αυτά τα σοβαρά θέματα τα οποία τίθενται. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, πρέπει να δω. Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσατε τώρα να αντιδράσετε στα όσα ακούσατε. Δεν νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτό που ακούσατε ήταν καινούριο για σας. Συνήθως αυτό το χρόνο κρατάμε 10 λεπτά, γιατί βλέπετε υπάρχουν και ευρωβουλευτές που θέλουν και αυτοί να σχολιάσουν και μετά τη συζήτηση σίγουρα θα μπορέσετε να έχετε και άλλο χρόνο εφόσον το επιθυμείτε. Πολύ καλά, κυρία Πρόεδρε, τότε ναι. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Τέσσερα κυρίως θέματα συζητήθηκαν εδώ την τελευταία μία ώρα περίπου. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο θέμα των ε, EDPs που είναι πιστεύω και εγώ το πιο ε, σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε σήμερα. Δυστυχώς θλίβαμε που το θέμα αυτό χρησιμοποιείται εδώ σήμερα σαν ε, ένα εργαλείο με χωρίς να δίνεται αρκετή προσοχή στο ίδιο το θέμα των μετατοπισμένων των προσφύγων. Ναι, σήμερα υπάρχουν ε, ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια της χώρας, γιατί αυτοί οι 280.000 που ήρθαν εκεί, μεταξύ αυτών κάπου 10.000 έχουν ήδη παραδεχτεί τις διασυνδέσεις τους με την τρομοκρατία βάσει πληροφοριών που έχουμε από αυτούς που έχουν συλληφθεί, που έχουν ε, μιλήσει για το κίνημα και που έχουν εντοπιστεί. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλοι. Θα σας διαβάσω μια ανακοίνωση που έγινε από τον Υπουργό στη Γενέβη πρόσφατα που αναφέρεται στις στατιστικές. Αλλά συγχρόνως θέλω να πω ότι περίπου το ένα έκτο των μετατοπιστέντων, των προσφύγων, έχουν ελευθερωθεί, έχουν αφαιθεί. Και κυρία Πρόεδρε, τέσσερις μήνες, μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που σταμάτησε η τρομοκρατία στη Σρι Οι πρόσφυγες αυτές δεν είναι ένα ασυνήθιστο φαινόμενο να ένα χάρτη εδώ που δείχνει τις διάφορες χώρες όπου υπάρχουν τέτοιοι πρόσφυγες. Και στο Αζερβαϊτζάν έχει 600.000. Η Γεωργία 300.000. Σε πολλές χώρες υπάρχουν. Γιατί εσείς παίρνετε την Σρι Λάνκα ενώ εμείς κάνουμε πολλή δουλειά. Όπως είπα και χτες, όταν ξεκίνησε η έκθεση για αυτό το θέμα, είναι πως βλέπει κανείς το θέμα. Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Για τη δουλειά που κάνουμε, είμαστε στη διαδικασία να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αφήνονται ελεύθεροι. Ορισμένοι έχουν επανακατασταθεί εκεί που έχουν εξουδετερωθεί οι νάρκες Άλλοι πάνε σπίτια τους, άλλοι πάνε στις οικογένειές τους. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλουν. Εκείνοι από τις 280.000, σας είπα ότι 10.000 έχουν ήδη πάρει ταυτότητες, 150.000 έχουν ελεγχθεί και έχουν αποδειχθεί αθώοι και δίνονται σε αυτούς διευκολύνσεις για να μπορέσουν να εγκαταλείψουν τους καταβλισμού. Είναι λάθος λοιπόν να λέτε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για αυτού τους ανθρώπους και ότι ζουν κάτω από κακές συνθήκες. Επίσης πρέπει να σας πω ότι 1236 ευθερώθηκαν πριν από ένα μήνα. Επίσης, ειλικρινά λυπάμαι για αυτά που λέτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πριν από λίγο μας ε, συνεχάρει για τα όσα κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί τότε αν ανησυχείτε για την κατάστασή τους. Οι διεθνείς οργανώσεις ζητήθηκαν να φροντίσουν να, επειδή υπήρχε θέμα ασφάλειας για αυτούς τους ανθρώπους, να βάλουμε έτσι να χτίσουμε δηλαδή τους καταβλισμούς αυτούς. Όμως το αρνήθηκαν οι οργανώσεις γιατί είπαν ότι αν γίνει αυτό θα είναι στο διενικέστα οι καταβλισμοί αυτοί, θα παραμένουν για πάντα. Και δεν έγινε. Το πάτωμα, να, να μπει στο πάτωμα, αντί να είναι χώμα, να βάλουμε τσιμέντο κάτω. Από το ICG ο υπεύθυνο είπε ότι κανείς δεν έχει πρόσβαση, ενώ αργότερα είπε όταν μιλάμε με τους ανθρώπους αυτούς. Το τελευταίο, το δεύτερο είναι αλήθεια. Ναι, 54 μη κυβερνητικέ οργανώσει και διεθνεί οργανώσει έχουν πρόσβαση στου καταβλισμού. Αλλιώ πώ λέτε ότι μιλάτε με αυτού του ανθρώπου, κυρία Πρόεδρε. Όσο για το μακροπρόθεσμο σχέδιό μα. Να, ο χάρτη που δείχνει τι περιοχέ στη Σρι Λάνκα για τις οποίες έχουμε αποφασίσει πού θα βγάλουμε τις νάρκες. Εδώ βλέπετε είναι που υπάρχουν οι μεγαλύτεροι καταβλισμοί ή οι πορτοκαλί. Οι... Και εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι όταν γυρνάνε στα σπίτια τους πρέπει να μπορούν και να καλλιεργήσουν και να τα πράσινα κομμάτια είναι εκεί που μπορούν να έχουν τις καλλιεργίες τους. Και ποιους ανθρώπους καταστούμε εκεί. Πολλοί. Το 96 ήρθαν σε αυτή την περιοχή. Είναι λοιπόν λογικό οι άνθρωποι που είναι από τη Ζιάφνα, ας πούμε και βρίσκονται τώρα στους καταβλισμούς θα πάνε πίσω. Αλλά μέχρι να πάνε εκεί για να χτίσουν τα σπίτια τους, ε ναι, βρίσκονται σε μια προσωρινή κατάσταση. Αλλά αυτά είναι γνωστά. Όταν David λέει ότι δεν γίνεται τίποτα, νομίζω ότι σφάλει. Το άλλο που θέλω να πω για, για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων θα επανέλθω μετά. Αλλά κάτι άλλο για την άμεση απελευθέρωση. Ο κύριος της Ανάγκαν. Είναι, ε, είναι φίλος. Κι εγώ είμαι δημοσιογράφος. Και ο Ντέβιτ και ο Σουνάντα είπανε είπε ότι ο δημοσιογράφος αυτός καταδικάστηκε σε καταναγκαστικά έργα επειδή έγραψε δύο άρθρα. Όχι, έγιναν δίκες, σωστές, 18 μήνες κράτησε η διαδικασία. Για τρία πράγματα. Το ένα ότι έγραψε τρία άρθρα. Αυτό ήταν μία από τις τρεις κατηγορίες και πήρε πέντε χρόνια για αυτή την ε, κατηγορία. Αλλά η άλλη κατηγορία ήταν ότι με τα άρθρα αυτά προσπαθούσε να δημιουργήσει ταραχές αλλά το τρίτο για το οποίο πήρε 10 χρόνια ήταν, ήταν θέμα οικονομικό χρημάτων που έπαιρνε από τους τρομοκράτες και αυτό αποδείχτηκε. Ο κύριος Τιζανάγκμαν διορθώνει μερικά πράγματα. Αυτό γιατί δεν το διορθώνει. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να λέτε ότι η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματο πρέπει να παραμείνει και μετά όταν έχετε ένα κακό αποτέλεσμα σε δίκη λέτε «Α, όχι, δεν είναι καλό». Ή το ένα ή το άλλο ισχύει. Το ίδιο δικαστικό σύστημα δίκασε και αυτούς που φύγαν από το Κολόμπο. Άρα δεν μπορείτε να αμφισβητείτε τη δικαστική εξουσία. Δεν λέω ότι η κυβέρνηση της Σρι δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν λέω ότι δεν έχουμε μπελάδες, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Τέλος. Θέλω να αναφερθώ και σε αυτά που είπε ο κύριο Τεσάμπρια που λέει ότι είναι εδώ γιατί είναι σε εξορία. Αυτό εξορία. Για έξι μήνες, γιατί απειλεί τη ζωή του. Ορίστε, διαβάζω εδώ κυρία Πρόεδρε, δήλωση του δόκτωρο Σπάρτος του που είναι εκτελεστικός διευθυντής ε, κέντρου που λέει ότι το 2008 ο κύριος ε, αυτός δέχεται την παρέτησή του από την Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης και που είχε από το 2002 διότι και συγχρόνω επέστρεψε όλα τα χρήματα στην οργάνωση μετά από έρευνα που έγινε για οικονομικέ ανομαλίε για ένα σχέδιο για το οποίο ήταν υπεύθυνο το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τι θα κάνει με την παρέτηση αυτή. Διαβάζω επίσης από άλλη εφημερίδα η ηγέτη του Σάντε που το 2009 το Μάιο έγραψε κατηγορείται για καταχρήσεις δημοσιογράφος παρετείται και δέχεται καταχρήσεις που έκανε σκάνδαλο ερευνείται για κατάχρηση ε, οικονομικών μέσων που δόθηκαν στο κινημάτο. Ορίστε, θα σας τα καταθέσω τα έγγραφα αυτά και σας τα λέω αυτά κυρία Πρόεδρε γιατί να, ποιος είναι αυτός ο οποίος ήρθε εδώ για να μιλήσει για την ελευθερία των μέσων. Ακριβώς εξαιτίας ανθρώπων σαν και αυτών που έχουν καταχραστεί το δικαίωμα εκπροσώπησης ε, ε, του κόσμου στα μέσα ενημέρωσης, γι' αυτό υπάρχει πλήγμα στην αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης σήμερα. Να, Επίσης θέλω να κάνω έκκληση σε εσά. Όταν φέρνετε ανθρώπους εδώ να μιλήσουν για τη Σρι Λάνκα, να φέρνετε καθαρούς μάρτυρες και όχι ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοια στην πλάτη του. Γιατί να. Ορίστε, ποιο σας είπε να τον φέρετε. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ότι τηρήσατε και τον χρόνο μιλία σας. Φυσικά σέβομαι το δικαίωμά σας να μιλήσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θέλουμε, θέλω να σέβομαι και το χρόνο μιλίας όλων των συναδέλφων. Έχουμε τον κύριο Μάρτιν και τον πρώτον ομιλητή εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για την ε, σαφή παρουσίαση που έκαναν. Έχω μια σαφή τώρα εικόνα της κατάστασης στη χώρα. Εμεί ω Κοινοβούλιο εκφράσαμε σοβαρέ ανησυχίε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πριν το τέλο του πολέμου, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, ψηφίσματα και κάναμε και μία ακρόαση τέλο Μαρτίου. Πριν τον πόλεμο, πριν το πέρα του πολέμου. Δεν χρειάζεται να σα θυμίσω. Το λέω καλύτερα για του φιλοξενμένου μα. Ω Επιτροπή, εμεί δεν μεροληπτούμε. Είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν παίρνουμε μέρο υπέρ των ταμίλη τη κυβέρνηση. Είμαι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε την αλήθεια και να βρούμε μια λύση για πρόοδο. Προσωπικά θεωρώ ότι η κυβέρνηση του Στριλάνκα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Αν ήθελα να δείξουν ανθρωπισμό και ταπεινοφροσύνη μετά την νίκη, θα έπρεπε να φροντίσουν για τη συμφιλίωση στη χώρα και συμφωνώ με του δύο μιλητέ μα που είπαν ότι οι Ταμίλ, όχι οι Ταμίλ Τάγκερ, μετά το πέρας της σύρεξης αυτής η συμπεριφορά τους της κυβέρνησης ουσιαστικά δημιουργεί νέα πηγή δυσπιστία και ενδεχομένως μελλοντική πηγή τρομοκρατών. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε γιατί ο πιο μεγάλος στρατολόγος για τους τρομοκτώπεδα αυτά τα IDPs ο πρέσβης Άκουσα με προσοχή τι είπε για ανεξάρτητου παρατηρητέ, αλλά από τα στοιχεία που εμεί έχουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τα Ηνωμένα Έθνη, η Ένωση, οποιαδήποτε άλλη οργάνωση να έχει πρόσβαση στα στρατόπεδα αυτά, να δει τι γίνεται εκεί. Αν τα πράγματα πάνε τόσο καλά στα στρατόπεδα, γιατί μας αρνούνται την πρόσβαση. Άρα έχουμε λόγους να δυσπιστούμε. και τους δίνουν άδειε στα άτομα να βγούνε και να γυρίσουν ακόμα και στις σπίτι τους. Άμα να γυρίσει κανείς στο σπίτι του και κινδυνεύει να πατήσει νάρκη, γιατί να γυρίσει. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα που δεν τηρούνται. Δεν έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να μετακινηθούν τα άτομα αυτά από τα στρατόπεδα να δουν κατά πώς συνδέονται με τους τίγρες του τα ή όχι. Δεν μιλάω για εθνοκάθαρση, αλλά σχεδόν περί αυτού πρόκειται. Όταν εκτοπίζονται άτομα από ένα μέρο τη χώρα σε άλλο, έτσι ώστε να μην εμφανιστεί ξανά πλειοψηφία του Ταμίλου στο Βορρά, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί είναι ελευθεροτυπία. Άκουσα τον πρεσβευτή, αλλά δεν πείθομαι. Και δεν νομίζω οι τόνοι στυλ ε, μακάρθι να βοηθάνε, να τον βοηθάνε. δεν ε, ε, βοηθάνε την εικόνα της κυβέρνησης. Τώρα γιατί ο gsp συν. Το είπα στην Επιτροπή Εμπορίου. Εμείς ως Ένωση καθυστερήσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, GSP GSP-SIN, Το γενικευμένο προτιμήσεων. Το δίνουμε σε χώρες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα έπρεπε να το είμαστε θέση να το άρουμε αν συμβαίνει το αντίθετο. Εγώ θεωρώ ότι μια χώρα της δίνεται αυτό το καθεστώς και αρνείται να συνεργαστεί με την Ένωση για έρευνα, αυτή η ίδια δίνει την αφορμή να της αποσυρθεί, να της αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα. Μέχρι ότου έχουμε αποδείξεις περί του εναντίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από ό,τι διαβάζουμε στον τύπο, και έχουμε δύο εκθέσεις και η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει δει την έκθεση αυτή, έχουν διαρρεύσει ορισμένα από τον τύπο. Η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Η έκθεση αυτή λοιπόν, από τα στοιχεία που έχει αυτή η έκθεση, μας υπαγορεύει οπωσδήποτε να αφαιρέσουμε αυτό το καθεστώς από τη Sri Lanka GSP sin Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάρτιν, η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο. Και εγώ για τους εσωτερικά ιδιωγμένους, τους IDPs, θα πω τα εξή. Ακούσαμε πολλές πληροφορίες από διάφορες πηγές, ακούσαμε και πιο λεπτομέρειες πληροφορίες μόλις τώρα από τον πρέσβη της Στριλάνκα. Ε, και νομίζω ε, πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι επίγον το να αναλυφθεί τώρα δράση καθώς πλησιάζει η εποχή των μουσώνων. Και γι' αυτό ίσως θα πρέπει η Επιτροπή μας να στραφεί στην κυβέρνηση της Στριλάκα και να αξιώσει ρητά τόσο η UNICEF όσο και η UNHCR δηλαδή είπατε αρμοστία του για τους πρόσφυγες να έχουν και πάλι πρόσβαση σε αυτά στα στρατόπεδα αυτού του καταβλισμού. Ε, ακούσαμε και πάλι από τον πρόσωπο τη Σριλάνκα ότι απελευθερώθηκαν άτομα. Οι Amnesty International μας είπαν ότι ναι, γύρω στα 8.000 άτομα, ιερείς, ε, δηλαδή τόσο Ινδουιστές ιερείς όσο και καθολικοί ιερείς απελευθερώθηκαν, αλλά υπάρχει η περίπτωση όπου αυτά τα άτομα δεν μπορούν να επιστρέψουν στις περιοχές όπου διέμεναν προηγουμένως. Και εδώ αναφέρονται ε, περιοχές υψής της ασφαλείας που κρατούνται από τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει κάποια δυνατότητα να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Ναι, είναι ένα πρώτο βήμα να απελευθερωθούν αυτά ε, τα άτομα τους ώστε να μπορέσουν να ε, διαμείνουν για παράδειγμα στις δυο θρησκευτικέ κοινότητες ενωρίες αλλά πρέπει και να ληφθεί και το δεύτερο βήμα δηλαδή να επιστρέψουν στις κατοικίες τους αυτά τα άτομα. Επίσης ακούσαμε ότι διώκονται πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και μάλιστα έχουν θανατωθεί πολλοί δημοσιογράφοι στη Σρι χωρίς να ασκούνται ποινικέ διώξεις. Ε, και όπως είπατε ε, και εσείς ε, Πρόεδρε χθες σε σχέση με την κατάσταση στη Ρωσία είναι παρόμοιο εδώ ε, το ζητούμενο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί το καθεστώς της ατιμορρησία. και εδώ θα πρέπει να ε, αξιώσουμε από την κυβέρνηση της Σρι να ξεκινήσει έρευνε ούτως ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο υπεύθυνο για την εκάστοτε δολοφονία. Και ίσως θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε εδώ στην επιστολή μας να ε, ανταποκριθεί και να συμμορφωθεί με τη δήλωση που είχε κάνει σχετικά με αυτά τα δικαιώματα η κυβέρνηση προς ε, τον πρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Και επειδή ακούσαμε κάποιες απόψεις εδώ, ε, θα πω ότι αυτό που είπε ο πρόσωπος του National Crisis Group είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μετά από αυτόν τον 30 ετή πόλεμο από τον οποίο έχουν υποφέρει όλοι και οι ε, και οι ε, να εντοπιστούν και εκείνοι οι οποίοι είναι πραγματικοί ε, συνεργάτες ε, των ομοκρατών, ώστε να απομονωθούν και να υπάρξει μια πραγματική λύση του προβλήματο που αποτέλεσε ευθύ εξ αρχή την αιτία αυτή τη διαμάχη. Δηλαδή, θα πρέπει να αντιληφθούμε εδώ ότι δεν θα πρέπει να είμαστε μονομερεί, θα πρέπει να επιτύχουμε το καλύτερο για του πολίτε ασχέτω του σε ποια εθνική ομάδα ανήκουν. Ευχαριστούμε την κυρία Λόχμιλα. και τα δύο ε, μέλη που πήραν το λόγο έκανα κάποιες ε, πολύ πρακτικές προτάσεις. Και η κυρία Λοχμιλέρ αναφέρθηκε ε, στο, στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Λάγκα και την ε, δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή κατοικίας για τα άτομα που φεύγουν από τους καταβλισμούς. Νομίζω πως θα ήταν σημαντικό τώρα να ακούσουμε κάποιες απόψεις από τους προσκαλεσμένους μας για τα όσα υπόθηκαν και στο τέλος να ακούσουμε και την άποψη του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα. γύρω στη μισή ώρα, εάν είναι όλοι σύντομε στι παρεμβάσει του. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Στρόλαν, μετά στη συνέχεια ο κύριο Δεσάμπλε και στη συνέχεια ο κύριο Σερά. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ναι, ε, άκουσα πως υπάρχει αρκετή ομοφωνία ε, στην αίθουσα, αλλά και γενικά σε όλο τον κόσμο, σε ό,τι αφορά το λόγο πρόβλημα των ιστορικά εκδοχημένων, των IDPs δηλαδή, αλλά σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία, ε, θα ήθελα να τονίσω, ε, κύριε Πρέσβη, αντί να αναφερθείτε στο ζήτημα της ελευθερίας του τύπου στη Στριλάνκα επιτεθήκατε σε έναν δημοσιογράφο που κατά κάποιο τρόπο αποδεικνύει ακριβώς αυτό που υποστήριζε εκείνο. Σε ό,τι αφορά όμως εσωτερικά και Ο πρέσβης ανέφερε πως το 1 έκτο έχει ήδη φύγει από αυτά τα τόπα, από του καταβλισμού. Είναι ενδιαφέρον αυτό το νούμερο, δεν το έχω δει πουθενά. Έχω εδώ ένα κατάλογο από όλε τι ε, αντικρουόμενε κιόλα δηλώσει τη κυβέρνηση, ε, και δεν υπάρχει ε, καμία δηλώση που να αναφέρεται στο 1 έκτο. Είναι κάτι καινούριο που ακούμε. Αν μπορείτε να μα το αποδείξετε κιόλα θα ήταν χρήσιμο, κάτι καινούριο και μετά μας λέτε ότι δεν επιτιθέμεθα στο Αζερμπαϊτζάν και στη Γεωργία. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για άτομα που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση από το 1994 και προφανώς επιτιθέμεθα αν χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση του πίκοντα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν, τη Δευτέρα θα δημοσιεύσουμε ε, ε, μια έκθεση ό,τι αφορά τον Αγκόνο Καραμπάχ και την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Και σα λέω από το 1994. Και δεν θέλουμε οι καταβλισμοί στη δική σας χώρα να υπάρχουν σε 15 χρόνια. Γιατί δεν θέλουμε έτσι Γιατί δεν θέλουμε να μονιμοποιηθούν αυτοί οι καταβλισμοί. Η διεθνή κοινότητα δεν επιθυμεί τη μονιμοποίηση αυτών των στρατοπέδων. Νομίζω πως αυτές είναι πολύ σαφές απαντήσεις στα όσα είπατε. Είπατε πως υπάρχουν κάποιες ε, ε, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση, ε, δηλαδή κάποια άδεια ε, δεν άκουσα ακριβώ το νούμερο. Μπορείτε να μου πείτε πιο συχνά ποιο είναι αυτό το νούμερο. Και αν πράγματι έχουν λάβει μια τέτοια άτομα. Γιατί τότε δεν μπορούν να φύγουν από αυτού του καταβλισμού τελικά, γιατί δεν μπορούν να πάνε σπίτια του, γιατί δεν μπορούν να δουν του ε, συγγενεί του, γιατί είναι φυλατισμένοι. Ε, και για να πω κάτι πως είπατε κάτι σε σχέση με αυτόν τον δημοσιογράφο ο οποίος καταχράστηκε το δικαίωμα του ελεύθερου λόγου από την πλευρά του, μα αυτό δεν είναι, κάτι, δεν είναι κατάχρηση ενός δικαιώματος, είναι δικαίωμα αυτό. Ο πρέσβης είπε κάτι εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Μπορεί αυτό η εξοχότητά σας να αναμένει λίγο. Ε, γιατί α, δεν ήσασταν στο μικρόφωνο και έτσι δεν μπορούσε να υπάρχει ερμηνεία. Ναι κυρία Πρόεδρε, δεν είπα κάτι τέτοιο σχέση με τον δημοσιογράφο. Δεν αναφέρθηκα στο ζήτημα του ότι εκφράζει γραπτός τις απόψεις του. Απλώς είπα πως ε, για παράδειγμα το άρθρο το οποίο ανέφερα αναφέρει πως ε, κάποιο χρηματοδοτούνταν από μια τρομοκρατική οργάνωση. Τι θα γινόταν εδώ, για παράδειγμα, αν γνωρίζετε πως κάποιος χρηματοδοτείται από την Αλκάιντα. Ναι, εάν χρειαστεί, θα σας δώσουμε χρόνο ομιλία στο τέλος. Αλλά με βάση τη σειρά ομιλητών που έχουμε, θα δώσουμε καταρχήν το λόγο στον κύριο Τεσάμπρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκαν ε, κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά ε, κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια που αποτελούν και το λόγο για τον οποίο δεν μπορούν να απελευθερωθούν κάποια εσωτερικά εκδιωγμένοι. Να πω πως ο πρώην ε, πρέσβης ε, στη Γενέβη από την πρώτη της Λάγκα είχε συμμετάσχει σε μια ειδική διάσκεψη που είχε λάβει χώρα το Μάιο στη Γενέβη ε, κατά του ε, ε, ε, ψηφίσματος το οποίο προετοιμαστεί το Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά ε, έχασε την θέση του δηλαδή δεν ήταν πλέον ο και την περασμένη εβδομάδα μας είπε 10 με 20.000 μπορεί να υπάρχουν οι οποίοι να έχουν απελευθερωθεί. Αλλά τι συμβαίνει με του υπόλοιπου 200 πρέπει να απελευθερωθούν. Αυτό δεν είναι δικά μου λόγια, είναι αυτά του πρώην πρέσβη τη Τριλάνκα Και για τον ελόγο δημοσιογράφου δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία. Καταδικάστηκα με βάση ένα ε, αντιτρομοκρατικό νόμο τον οποίο έχει εγκρίνει ο ίδιος ε, ο κύριος Ρατζαπάξα α, ως ε, τέτοιον, ως ο ίδιος δηλαδή ο τωρινός ε, πρόεδρος στο παρελθόν είχε καταφερθεί εναντίον αυτού του νόμου, ότι είναι αντιδημοκρατικός ο οποίο θεωρεί πω οι ομολογίε αποτελούν αποδεκτικά στοιχεία. Δεν υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία ότι χρηματοδοτήθηκε από του Tamil Tigers, πέρα από την ομολογία. 1.005 δολάρια. Όχι 10.000 δολάρια που αναφέρεται. Και γιατί χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα. Η κυβέρνηση είπε ότι ε, ε, αξιοποίησε αυτά τα ε, χρήματα για να εκτυπώσει τα δύο άρθρα του. Δηλαδή καταδικάστηκε ότι έλαβε χρήματα από τους Tamil Tigers για να τυπώσει τα άρθρα του. Έλαβε λοιπόν τα χρήματα όχι για να διακηρύξει την ένοπλη βία, για να ε, ε, πολεμήσει εναντίον της κυβέρνησης οτιδήποτε άλλο, για να συγγράψει και να εκτυπώσει τα άρθρα του. Και στα σχετικά σχόλια που είχε κάνει εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην, ε, στο σταθμό Αλτζαζίρα, το είχε πει ότι ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ότι πράγματι καταδικάστηκε για αυτό το λόγο, για αυτά τα δύο άρθρα. 10 συν 10 χρόνια, 20 χρόνια συνολικά. Είκοσι λοιπόν χρόνια καταδίκης για τη συγγραφή δύο και μόνο άρθρων. Και σας λέω πρώην ε, ε, ηγέτες των Tamil Tigers ε, που ήταν αρμόδιοι ουσίων αστυνομικών κατά τη δεκαετία του 1990 έχουν καταλάβει τώρα θέσεις υπουργών στην κυβέρνηση είναι λοιπόν μια πολιτική δίκη αυτή που έλαβε χώρα για να δοθεί το μήνυμα σε άλλους ότι αν γράψετε τέτοια άρθρα αυτό θα πάθετε. Αυτά τα άρθρα γράφτηκαν το 2004. Τίποτα δεν συνέβη με βάση αυτά τα άρθρα. Και δύο σύμβουλοι της κυβέρνησης ε, είπαν, κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι αυτά τα άρθρα δεν αποτελούν, ε, δεν προξενούν ε, βία. Δεν καλούν κανένα στο να προσφύγει στη βία. Άρα λοιπόν το να μας λένε ότι εδώ ακολουθήθηκαν κανονικέ διαδικασίες δεν είναι σωστά. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των εσωτερικών εκδιωγμένων, υπήρξε μια νέα ενημέρωση από τον ειδικό α, διευθυντή της αστυνομία, που είπε το εξή. 20.000 IDPs, εσωτερικά εκδιωγμένοι, διέφυγαν από τους καταβλισμούς. Ποιος είναι υπεύθυνο για αυτό μα λένε ότι έπρεπε να του απελευθερώσουν επειδή υπάρχουν ανησυχίε σε ό,τι αφορά την ασφάλειά του. Πώ λοιπόν επέτρεψαν να, να, να, να διαφύγουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Και σα λέω πω το παραδέχτηκαν αυτό οι ειδικέ δυνάμει τη αστυνομία, δεν το λέω εγώ. Και το, και το ανέφερε στην εφημερίδα Island, η οποία δεν είναι μια αντικυβερνητική εφημερίδα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι φτωχοί. Έχουν ε, καταθέσει 500 εκατομμυρίων ρουμιών στις τράπεζες. «21.000 λογαριασμοί έχουν ανοιχθεί μέσα στους τους, ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους και να μαγειρεύουν ε, το φαγητό τους. Ε, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια χρήματα, μπορούν να επιστρέψουν στις δικές τους κατοικίες, μπορούν να εργαστούν και μπορούν να μεταβούν για να νοικιάσουν μια κατοικία γιατί λαμβάνουν και βοήθεια από τις οικογένειε του. Άρα λοιπόν 500 εκατομμύρια ρούπια έχουν καταθέσει, οπότε δεν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι. Δεν έχουμε αυτού του λόγου ασφαλεία, για παράδειγμα, μα λένε ε, ότι υπάρχουν άρκε και γι' αυτό ανησυχούν. Αν αυτό ισχύει, τότε γιατί δεν έχουμε πρόσβαση όλοι μέσα σε αυτού του καταβλισμού. Προκαλώ την κυβέρνηση να αποδείξει επίση να μου πει ε, πού είναι τα χρήματα αυτά τα οποία εγώ υποτίθεται πως υπεξαίρεσα. Εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, γιατί δεν μου τα δείχνει κανένας, δεν υπάρχουν πουθενά. Εάν θέλετε μπορώ να σας ε, αναφέρω εγώ να σας παραπέμπτω σε εκατοντάδες άρθρα. Αυτές οι εφημερίδες ε, μπορούν να λένε οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορούν να αναφέρονται σε κάτι εφημερίδες το οποίο τελικά δεν έχει αποδειχθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Εγώ απλά θέλω μια επιδικοδομητική συζήτηση. Έχουμε, συζήτη, έχουμε συναντήσει τον Πρόεδρο, έχουμε συναντήσει εκπροσώπου τη κυβέρνηση και θα πρέπει να επιτύχουμε πρόοδο σε αυτή την ε, χώρα. Και αν θέλουμε πρόοδο, θέλουμε συμφιλίωση, όχι να κατηγορούμε ο ένα τον άλλον. Γι' αυτό και εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Εάν θέλετε να προοδεύσουμε, πρέπει να δούμε ποιο δολοφόνησε δημοσιογράφου, τι μπορούμε να διορθώσουμε, ποιο είναι ο τρόπο μπροστά. Αυτό ζητώ από την ε, κυβέρνηση. Και αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, χρειαζόμαστε συμφιλίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δεσάρκλια, για τα όσα μας είπατε. Ο κύριος Τζεράρ, θέλετε και εσείς να σχολιάσετε. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Ίσως το μεγαλύτερο φόρουμ στην 64η συνέλευση είχε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό της Λάνκα, που είπε μια από τις κύριες προτεραιότητές μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανθρωπιστικές ανάγκες των μετατοπισμένων και να διασφαλίσουμε την ε, αξιοπρεπή επιστροφή τους στα σπίτια τους, την ευημερία τους που, βρίσκεται σε, που οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε μεταβατική ε, περίοδο και θέλουμε να δεχτούμε για αυτού διεθνεί προδιαγραφές. Η Σρι Λάνκα θέλει να συμμορφωθεί με τις διεθνείς τη υποχρέωσει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικών προδιαγραφών. Τέτοιου είδου δηλώσεις μας αρέσουν πάρα πολύ. Αναλαμβάνουν μια υποχρέωση. Και είναι ξεκάθαρο ότι εμεί αυτό που θέλουμε από την κυβέρνηση τη Σρι Λάγκα είναι να εξακολουθεί τι προσπαθίε τη για να εφαρμόζει το διεθνέ δίκαιο και τους ανθρωπιστικούς κανόνες. Για το θέμα τώρα των καταβλισμών, που από ό,τι φαίνεται είναι αμφιλεγόμενο με ποιο τρόπο το χειρίζονται. Εμείς ξέρουμε ότι εξορισμού αυτοί οι καταβλισμοί είναι προσωρινοί. Είναι για πολίτες και από τη φύση τους πρέπει να είναι προσωρινοί. Η εμπειρία μου βέβαια τα τελευταία 17 χρόνια είναι ότι στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές όπου υπάρχουν τέτοιοι καταβλισμοί και έχω πάει σε τόσο πολλά μέρη, πάντα επιμένουμε για το προσωρινό των καταβλισμών, όχι μόνο επειδή από τη φύση τους πρέπει να είναι τέτοια, αλλά και γιατί καλύπτουν ε, το στόχο τους. Προστατεύουν τον κόσμο για το χρόνο που πρέπει να τον προστατεύσουν. Υπάρχουν ε, οι αρχές, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για τους μετατοπισμένους. Αυτό είναι ένα εργαλείο που το έχουμε στη διάθεσή μας από το 1998 και πολλές χώρες έχουν συνυπογράψει και η Σρι Λάγκα επίσης. Έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες για να το αντιλαμβάνονται και όλες οι πλευρές μέσα στη Σρι Λάγκα. Και γι' αυτό και θέλουμε η ανθρωπιστική κοινότητα αλλά και όλοι οι υπόλοιποι να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήρες αυτές γραμμές και βέβαια και η κυβέρνηση της Σριλάνκα. Το τελευταίο που θέλω να θέξω είναι το εξή. Είμαι σίγουρη ότι και άλλοι και οι Κομισιόν θα συμφωνήσουν μαζί μου για το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δουλεύεις για ανθρωπιστική βοήθεια να βρίσκεσαι σε τέτοια ατμόσφαιρα, σε τέτοιο περιβάλλον, σε καθημερινή βάση να μην ξέρει, αν θα έχει το δικαίωμα ή δεν θα έχει το δικαίωμα να μπει μέσα στο καταβλισμό. Να σε ελέγχουν επειδή κάνει ανθρωπιστικό έργο και να μην είσαι σίγουρος για το ότι η δουλειά που κάνει θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αξιοπρεπώς. Έτσι λοιπόν όλοι όσοι προσφέρουν τέτοια ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημα. Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μια τέτοια κατάσταση θα πάυσει προκειμένου αυτό το ηθικό τελικά δίλημα να μην υπάρχει πια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν είναι αποδεκτή μια τέτοια κατάσταση. Η κυβέρνηση της Σρι πρέπει να τηρεί τις υποχρώσεις της απέναντι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις προκειμένου αυτές να μπορούν να δουλέψουν. Πολλοί που συνελήφθηκαν πριν από μερικούς μήνες παραμένουν σε κράτηση. Υπάρχει μια κατάσταση όπου ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αντιδράσει έντονα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να προσθέσει έτσι καλώς πρέπει να πούμε εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπουμε εμείς τα πράγματα, υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα με τον τύπο στη Σρι Λάνκα. Γιατί ακούμε για έγγραφα τα οποία θα έπρεπε να δημοσιευθούν, αλλά δεν δημοσιεύονται, δεν δημοσιοποιούνται. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια δυσκολία. Να ξέρετε ότι Μόνο θετικές μπορεί να είναι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ ανθρώπων που έχουν εμπιστοσύνη μεν στους δε. Οπότε ευχαριστώ τον κύριο Τύρ ε, για όσα μας είπε από την Επιτροπή και ίσως θέλει ακόμα κάτι να προσθέσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, όπως και ο συνάδελφος, είπε έτσι και εγώ θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει απόλυτα την άμεση απελευθέρωση τουλάχιστον των περισσότερων μετατοπισμένων που βρίσκονται στους καταβλισμούς αυτούς όπως επίσης και την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων εκεί. Επίσης, Ξέρουμε ότι δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις ανθρωπιστικές μας απασχολούν με εξοδικαστικές ε, δολοφονίες, με απαχθέντες, με προβλήματα κυκλοφορίας πληροφοριών, ενημέρωσης και αλλού στη Σρι Λάγκα. Η Ερευνητική Επιτροπή που ορίστηκε από τον πρόεδρο της Σρι Λάγκα το 2006 σταμάτησε τις εργασίες της. Η εντολή της δηλαδή δεν παρατάθηκε. Η Ερευνητική αυτή Επιτροπή δεν δημοσίευσε συμπεράσματα και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οι εργαζόμενες στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, κάποιοι μάλλον από αυτούς, έχουν χάσει τη ζωή τους στην Σρι έχουν δολοφονηθεί και θέλαμε έρευνα προκειμένου να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Καταδικάζουμε φυσικά τις ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης που εξακολουθούν να ισχύουν. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να δουλεύουν ανεξάρτητα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό αναφέρεται στο καταστατικό τους έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα η κατάσταση των μετατοπισμένων είναι πιο κρίσιμη και πιο άμεση. Όμως πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι οι ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ευρύτερε. Δεν καλύπτουν μόνο τους μετατοπισμένους. Ελπίζουμε τώρα που ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε να υπάρξει αποκατάσταση. Και ελπίζουμε η Σρι να μπορέσει να κάνει κάτι όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όμως θέλω βέβαια να δώσω το λόγο και στους συναδέρφους εδώ για να κάνουν κάποια σχόλια. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε κύριε Τύρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ναι, θα είμαι σύντομος. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος. Άκουσα τον καλό μου φίλο, τον πρέσβη. Και έτσι εδώ πρέπει να σκεφτώ το εξή. Αν όλοι αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε για τα γεγονότα, θα προσπαθούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δεύτερον, δεν είπα ότι δεν γίνεται τίποτα για τους καταβλισμούς. Ούτε υπονόησα ότι είναι εύκολο να ασχοληθεί κανείς με τόσο πολλούς ανθρώπους, αλλά όπως τονίσανε εδώ και άλλοι, γιατί να πρέπει να ασχοληθούμε με τόσους πολλούς ανθρώπους και δεν τους αφήνουμε να φύγουν. Τα προβλήματα που έχουμε δει είναι τα εξή. Πρώτον, ορισμένοι όντως έχουν βγει από αυτούς τους καταβλισμούς, αλλά δεν έχουν ελευθερωθεί, έχουν μεταφερθεί σε άλλους καταβλισμούς κάποιοι. Έπειτα, έρχεται ο χειμώνα. Και είναι μια μεγάλη μα ανησυχία αυτή για το τι συνθήκε θα επικρατήσουν εκεί. Τρίτον, δεν υπάρχουν ε, ε, νάρκες σε όλες τις περιοχές από όπου προέρχονται αυτοί οι μετατοπισμένοι, ορισμένοι θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έπειτα, εμείς δεν έχουμε ακούσει να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα πρόσβασης και σε χώρες όπως το Αζερβαϊτζάν για παράδειγμα ή η Γεωργία όπου αναφερθήκατε εσείς ή την πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή του ΟΗΕ αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε είναι να στηρίξει η κυβέρνηση της Ριλάνκα, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τον ΟΗΕ και να μας επιτρέψει να βάλουμε σε εφαρμογή τα προγράμματα μας, τα ανθρωπιστικά, υπέρ αυτών των ανθρώπων. Εσείς πρέπει να μας βοηθήσετε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα και να μπορέσουν ελεύθερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τέλος, για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να επαναλάβω όσα έχουν αναφερθεί στον τύπο μέχρι τώρα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πάνω από 30 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί τα τελευταία 4 χρόνια, κάπου 70 είναι σε εξορία, όπως ξέρω εγώ. Και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιογράφων σε τέτοιες καταστάσεις που έχουμε από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα μας είπε. και για, τα... την ενημέρωσή τους γενικότερα. Περιμένουμε τη δημοσίευση της εκθεσής σας. Τώρα, τώρα. Για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της τόσο ενδιαφέρουσα ακρόασης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά όλους που ήρθατε εδώ, που μας ενημερώσατε για τα όσα ξέρετε εσείς για την ε, κατάσταση αυτή. Α, ο πρέσβης. Ναι, αλλά να είσαστε πάρα πολύ σύντομος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ασχοληθεί και με τα μέσα ενημέρωση και με του μετατοπισμένου. σας τα είπα αυτά. Δεν χρειάζεται να σας τα επαναλάβω. Ένα πράγμα θα πω μόνο για τους μετατοπισμένους. Σας έδωσα τα γραφό, κυρία Πρόεδρε και έχω και αντίγραφα τα οποία κυκλοφορούν στους ευρωβουλευτές εδώ. Που δίνουν τα στατιστικά δεδομένα. ανησύχησα ακούγοντας τον κόσμο εδώ με κάθε σεβασμό προς τους ευρωβουλευτές. Αφήστε τους να φύγουν και αν πέσουν σε και σας πέσουν. Με τι είναι αυτά. Τι ξέρω, εσείς στις χώρες σας μπορεί έτσι να τα κάνετε. Εμείς στη Σελέγκα δεν κάνουμε έτσι τα πράγματα. Νιώθουμε υπεύθυνοι για τους ανθρώπους μας. Είναι δικοί μας άνθρωποι και δεν θα τους αφήσουμε επειδή εσείς θέλετε. Όχι. Εμείς θα κάνουμε ότι είναι καλύτερο για τον κόσμο μας. Οι άνθρωποι αυτοί 30 χρόνια ε, τους ε, έχουμε υπόψη μας, πρέπει να, να μας δώσετε και εμάς, ε, να μας θεωρήσετε αθώους μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή μας. Μην μας λέτε πριν από τόσα χρόνια έγινε αυτό το δεύτερο, ο κύριος της Απρίας παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα λογική, αλλά αποδεικνύει αυτό ακριβώς που είπα ότι δηλαδή ο κύριος Τεζανάγραμ πήρε μόνο 1.500 δολάρια. Ο κύριος ε, Τεσαπριέλ επίσης έχει την τάση, όχι σύμφωνα με μένα, αλλά με τη χειρογράψη εφημερίδες. Αυτό όμως που πιο πολύ με ξέπληξε είναι Εντάξει, άρθρα λέτε, εφημερίδε, μάλιστα. Αν κάποιο γράψει ένα άρθρο κατά του συμμετισμού, εσεί τι θα κάνετε. Κάτι ακόμα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα σε δύο λεπτά να ολοκληρώσετε, γιατί και εγώ έχω να κάνω κάποια σχόλια. Θα ήθελα και εγώ δύο λεπτά. Πέντε λεπτά. Λυπάμαι. Όχι. Ωραία, ωραία. Ανθρώπινα δικαιώματα. Θα τα αφήσω και θα σας στείλω ένα σημείωμα για αυτά ώστε να ενημερωθείτε. Θέλω να αναφερθώ τώρα στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Εδώ δόθηκε εντύπωση ότι η κυβέρνηση της Σριλάνκα δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ε, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ξεκαθαρίζω σε εσά ότι η κυβέρνηση της Σριλάνκα δεν συμμετείχε στην έρευνα αυτή για θέμα αρχής. Και οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν. Και τι κάνουμε, είπαμε δεν θα συμμετάσχουμε στην έρευνα αυτή, είπαμε όμως ότι θα ασχοληθούμε με τις τρεις συμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε. Είχε δύο συναντήσεις στις Βρυξέλλες και στο Κολόμβο για το GSP και εμείς να, θα σας δώσω αυτό το αντίγραφο κυρία Πρόεδρε. Ed Memoir που καλύπτει όλες τις πλευρές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς κοιτάζουμε το θέμα του GSP Plus και έχουμε τα σχόλιά μας. Ο Υπουργός ετοιμάζει έκθεση για να απαντήσει στους εμπειρογνώμονες και λυπάμαι που σας απογοητεύουμε, μάλλον αυτό ακούσαμε πριν, όχι. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Εμείς θα ασχοληθούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιστεύουμε ότι όταν ε, εφαρμόζεται αποτελεσματικά, τι σημαίνει αυτό, 40%, 50%, 80%, 90%, 99%. Ποτέ κανείς δεν έχει ερευνήσει πλήρω το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι δεν υπάρχει κατόφλι, δεν υπάρχει όριο. Όσο μας αφορά λοιπόν, και η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει αυτό, αποφασίσαμε από πλευράς αρχής για το ότι η κυβέρνηση της Ριλάνκα θα συνεχίσει συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα που εκφράζει ως ανησυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε πάρουμε το GSP είτε όχι, εμείς θα φροντίσουμε να διορθώσουμε ό,τι εντοπίσουμε σαν πρόβλημα, γιατί ούτε εμείς είμαστε τέλειοι, όπως τέλειος δεν είναι κανείς. Και το αναγνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό και την τελευταία εβδομάδα εδώ, εκπρόσωπος εδώ τι λέει, λέει πρόσβαση σε 10 μέρες των εκπροσώπων του ΟΗΕ. Πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, εν κατακλείδη. Όσο η Επιτροπή αυτή και αυτό το Κοινοβούλιο σέβεται την Σρι με τον ίδιο τρόπο που εμείς σεβόμαστε εσάς, τότε θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστούμε πολύ που, κυρία Πρόεδρε, που δώσατε, στην ευκαιρία, που δώσατε την ευκαιρία αυτή στην κυβέρνηση της Σρι Έχουμε σαφή πληροφόρηση και το κάνουμε πώς να κρίνουμε την κατάσταση από εδώ και μπρο, και από όπου ακούσαμε ότι η Κομισιόν περιμένει από την Σρι Λάγκα να φροντίσει να πάψει αυτή η συνεχής κράτηση των εκτοπισμένων. Επίσης πρέπει να ε, συζητηθεί το θέμα της ατιμορρησίας και να το κράτος δικαίου να γίνει πραγματικότητα. Επίσης το θέμα της ελευθεροτυπίας είναι σημαντικά Ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα αυτό σε πολλές χώρες στον κόσμο όπου πρέπει να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν το δικαίωμα, που δεν τους επιτρέπεται μάλλον ελεύθερα να γράφουν και να δημοσιεύουν. Οπότε και η πληροφόρηση αυτή δεν περνάει στο, σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κύριε Πρεσβευτά, φυσικά στην Επιτροπή μας κοιτάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλε τι χώρε γιατί η Ένωση έχει εξωτερικέ σχέσει με όλε τι χώρε. Σας διαβεβαιώνω, θα υπάρξει ευκαιρία για μα να συζητήσουμε την ευκαιρία των εκτοπισμένων και στο Αζερβαϊζάν και στην Γεωργία. Απλώ δεν ήταν σήμερα στην εμερήσια διάταξη. Απαντώ εκ μέρου του συναδέλφου David Μάρτιν. Ξέρετε, ο κύριο Μάρτιν δεν είπε ότι ο κόσμο οι άνθρωποι θα πρέπει να αφαιθούν στο έλεος των ε, ναρκών. Φυσικά δεν εννοούσε αυτό. Αυτό που όλοι λέμε και νιώθουμε είναι ότι η κυβέρνησή σας χρησιμοποιεί το θέμα αυτό ως δικαιολογία για να μην κάνει τίποτα για τους εκτοπισμένους. Τέλος, θα ήθελα η κυβέρνησή σας να πάρει στα σοβαρά την ε, οδηγίες του ειδικού απεσταλμένου των ΗΕ Εθνών όσον αφορά τις απαιτήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα και όταν προσπαθείτε να καταπολεμήσετε τους ε, τρομοκράτες. Όλοι είμαστε κατά της τρομοκρατίας, αλλά δεν επιτρέπεται αυτό να γίνεται σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστούμε για τις μαρτυρίες σας. Όλα αυτά ήταν χρήσιμα για το Κοινοβούλιο. Θα εξακολουθούμε να συζητάμε και με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν για το θέμα των εγκεκριμένων προτιμήσεων. Σας ΕΕ. Ευχαριστώ. Μία διακοπή πέντε λεπτών και μετά το διαβριμένο Προεδρείο.